Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να ξεκινήσουμε. Και σας ζητώ συγγνώμη για αυτή την μικρή καθυστέρηση, γιατί δεν συνηθίζουμε να συνεδριάζουμε σε αυτή την αίθουσα. Άλλωστε η πρόσβαση στο κτίριο αυτό είναι πιο πολύ δύσκολη. C'est une réunion λόγω του χρονοδιαγράμματος είναι κάπως ασυνήθιστη αυτή η συνεδρίαση, γιατί έχουμε μόνο μισή μέρα, σε μια εβδομάδα μάλιστα που κανονικά είναι αφιερωμένη στις συνεδριάσεις των ομάδων, κάτι που περιπλέκει τα πράγματα και που εξηγεί την απουσία του μεγαλύτερου τμήματος των σοσιαλιστών. Βέβαια, έτσι εξυπηρετούμαστε για να έχουμε περισσότερες ψήφους εμείς, αλλά δεν είναι και πολύ ευχάριστη αυτή η κατάσταση ούτε από πολιτική άποψη, ούτε από οργανωτική, δηλαδή για το πώς θα οργανώσουμε τη, τη ζωή μας και τα προγράμματά μας. Ελπίζω στο μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών μας να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις που ούτε τις ψηφοφορίες διευκολύνουν ούτε την αποτελεσματικότητα των εργασιών μας εξυπηρετούν. Θα κοιτάξετε την σε διάταξη. Ο κύριος Αλφόνση προεδρεύει σε συνεδρία σε άλλη επιτροπή, και ζήτησε να αναβάλουμε το σημείο 7, τα σημεία 6 και 7, για τα δύο πρωτόκολλα με τρίτες χώρες για αλληλευτικά ζητήματα. Είχαμε προβλέψει ανταλλαγή απόψεων, αλλά όχι ψηφοφορία. Οπότε τα σημεία 6 και 7 αναβάλλονται για άλλη συνεδρίαση. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Σημείο 2. Ανακοινώσει του Προέδρου θα τις δείτε στο Κόμπου News. Δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω. Έχουμε την ομάδα παρακολούθησης για, τις για την κατηγορία 1β του προϋπολογισμού. 20 Απριλίου, συνεδρίαση. Ξέρετε τι είναι αυτά, αυτές οι ομάδες παρακολούθησης. Ο James Ellis. Ναι. Γνωρίζουμε τι σημαίνει monitoring groups, αλλά αντί να τους έχουμε ξεχωριστά κάθε φορά, δεν μπορούμε να έχουμε ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα για να μπορούμε να παρακολουθούμε και τις εργασίες αυτών των ομάδων παρακολούθησης. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το εγχείρημα και καλό είναι να έχουμε χρόνο να το παρακολουθήσουμε. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τα προγράμματα. Όντως, έβλεπα το αίτημα και μετά την πρωινή μας συνεδρίαση θα συνεδριάσουμε οι συντονιστές. Εκεί θα προτείνω ένα χρονοδιάγραμμα για το σύνολο των συνεδριάσεων και από τη στιγμή που θα το εγκρίνουμε οι συντονιστές θα σας το αποστείλουμε και σε αυτό το χρονοδιάγραμμα, όπως ζήτησε ο James Ellis. Έχετε και τις γλώσσες διερμηνίας, γίνεται και αναμετάδοση από το web stream στο κανάλι του Κοινοβουλίου και έχουμε πολλές ε, πηγές ενημέρωσης για, τον, για την έγκριση του προπολογισμού του 2010. Σε ό,τι αφορά την έγκριση των πρακτικών της 3ης Μαρτίου του 2011, αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις μέχρι το πέρα συνεδρίασης, θα θεωρήσουμε ως ε, συγκεκριμένα τα πρακτικά. Και περνάμε στην σειρά των σημείων της ημερήσιας διάταξης. Ίγκε Γκρέσλε... Πού είναι? Α, μπροστά μου ακριβώς. Είχα τυφλωθεί από τη λάμψη και δεν την είδα καν. Έτοιμα λοιπόν της κυρίας Γκρέσλε και της Έργα Τρίπελ να διεκπαιρεώσουμε εντάχει τα δικά του σημεία, γιατί έχουν και άλλες συνεδριάσεις μετά, οπότε Πρώτα θα ξεκινήσουμε με το σημείο 5 και 14 και μετά θα περάσουμε στο 4. Και θα τηρήσουμε αυστηρά το χρόνο για το κάθε σημείο. Η σε κάθε συνεδρίαση μας ενημερώνει για το, την πορεία των εργασιών για το δημοσιονομικό κανονισμό. Ευχαριστώ αγαπητέ Αλά. Έχω μια καλή είδηση και μια άσχημη. Η καλή είδηση είναι ότι έχει πλέον ολοκληρωθεί η έκθεση, έχει και 130 περίπου τροπολογίες και μόλις η γραμματεία θα έχει εξετάσει τις τροπολογίες και θα τις διανύμει. Η έκθεση είναι στα αγγλικά με λίγες ε, τροπολογίες και της Κιεθρό Μάιερ που είναι αρμόδια για τα κτίρια στα γερμανικά, άρα μπορεί κανείς να διαβάσει αμέσως την έκθεση. Και όλες οι συνάδελφοι και όλοι οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για το θέμα, ας εξετάσουν την έκθεση αμέσως. Την γράψαμε επίτηδε στα αγγλικά, ώστε να μπορούμε αμέσως να αρχίσουμε τις συζητήσεις. Η ομάδα εργασίας μας θα συναντηθεί ξανά την επόμενη εβδομάδα, όπου θα διεξέλθουμε την έκθεση άρθρο προς άρθρο και τροπολογία προς τροπολογία. Γι' αυτό νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα που είχαμε κάποτε υποβάλει μετά από επιθυμία των συντονιστών. Θεωρώ λοιπόν ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό εξακολουθεί να είναι εφικτό και γι' αυτό δεν κατανοώ και την επιστολή της Επιτροπής ε, ε, Ρέγγι, δηλαδή της Περιφερειακής Επιτροπής, που λέει ότι δεν γνωρίζει αρκετά πράγματα. Ο εισηγητής της Περιφερειακής Επιτροπής, που είναι και μέλος της ε, ομάδας εργασίας μας και έχει επομένω πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και μάλιστα και στο επίπεδο τη κοινοβουλευτική μας ομάδας έχω επαφή μαζί του σε άλλη ομάδα εργασία. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Όλοι α αρχίσουν την εργασία. Έχει μάλιστα και η Επιτροπή φτιάξει και μια homepage όπου είναι διαθέσιμα όλα τα έγγραφα. Άλλωστε τα, τα διαβιβάζουμε τα έγγραφα. Πάντοτε όλα αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ και ε, μήνες. Νομίζω λοιπόν ότι Ήδη εργαζόμαστε με μεγάλη διαφάνεια γιατί θέλω πολλοί να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Εγώ συλλέγω το Συμβούλιο, διότι εκεί είναι μόνο 27 μέλη και η Προεδρία έχει συγκεκριμένους συνομιλητές και έτσι μπορεί να προχωρεί. Το ΔΕ Συμβούλιο ήδη θα υποβάλει πρόταση της Προεδρίας του τούτη την εβδομάδα. Έχει λοιπόν ε, ολοκληρώσει την εργασία του σε αυτό το επίπεδο Προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε και ορισμένα πράγματα στην έκθεση, αλλά δεν θα ήταν σκόπιμο να την παραφορτώσουμε την έκθεση, γιατί αποδυναμώνουμε, αποδυναμώνουμε έτσι την διαπραγματευτική μας θέση. Ας αφήσουμε ορισμένα πράγματα λοιπόν. Θέλουμε αρκετά άλλωστε. Τώρα, η άσχημη είδηση είναι και πραγματικά τώρα πρέπει να ρηχτούμε στη δουλειά, πρέπει να διαβάσουμε πολλά κείμενα είναι άλλωστε πολύ περίπλοκη και δύσκολη εργασία αυτή, διότι το κείμενο στα τμήματα του που είναι σημαντικά για τα PPP, Financial Instrument, Shared Management, έχει τροποποιηθεί. Σήμερα θέλω να μιλήσω για ένα πράγμα που είναι σημαντικό για το Κοινοβουλίο, δηλαδή τις κατανάθεση πράξη, της Delegated Acts. Εμείς στην έκθεσή μας θα φροντίσουμε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Εκεί είναι και το σημαντικότερο θέμα μας, διότι εκεί πρέπει εμείς να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας, οι άλλοι δεν θα το πράξουν. Η βάση είναι το άρθρο 219 της ε, συνθήκης, όπου λέει ότι οι πράξεις αυτές μπορούν να μεταφερθούν στην Επιτροπή, δηλαδή νομικές πράξεις χωρίς χαρακτήρα νόμου, που να μην είναι ουσιώδη. οι διατάξει αυτέ να μην είναι ουσιώδη. Ωστόσο, το πεδίο εφαρμογή και η διάρκεια πρέπει να είναι σαφώ καθορισμένα. Και οι συνθήκε υπό τι οποίε εκδίδονται οι πράξεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται στον ίδιο τον κανονισμό. Εδώ υπάρχουν εξή δυνατότητε. Κοινοβούλιο και Συμβούλιο μπορούν να αποφασίσουν να ανακαλέσουν την ανάθεση αλλά η κατανάθεση πράξη μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνο εάν δεν ε, προβάλλει ενστάσει στο Κοινοβούλιο το συμβουλίου μέσα σε μια συγκεκριμένη προθεσμία. Αυτά τα περιλάβαμε εμεί στην νομοθετική πράξη. Έχουμε ήδη μια έκθεση πρωτοβουλία, την έκθεση Σάιερ για τι κατανάθεση πράξη, που η έκθεση αυτή προβαίνει σε μια ερμηνεία της συνθήκης όπου μάλιστα την συζητήσαμε και με την νομική υπηρεσία. Η έκθεση Σάιερ λέει σύμφωνα με την συνθήκη σε κάθε βασικό νομοθέτημα πρέπει να καθορίζονται οι εκμεταφοράς αρμοδιότητες αλλά πρέπει να λεχθεί και ποιοι είναι οι μηχανισμοί ελέγχου. Μετά η έκθεση Σάιερ η οποία μάλιστα εγκρίθηκε με 590 ψήφους πλειοψηφία ότι οι περιπτώσεις ανάκλησης έχουν, έχουν χαρακτήρα μόνο παραδείγματος αυτές που αναφέρονται στη συνθήκη. Και αυτό είναι το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε, δηλαδή κατά πόσον, μέχρι πού θέλουμε να φτάσουμε. Βλέπει μια δυνατότητα λοιπόν η έκθεση Σάιερ σε συμφωνία και με την νομική επιτροπή, αλλά δεν έχει ερωτηθεί η νομική υπηρεσία. Το ψάξαμε αυτό. Μέχρι πού θέλουμε να φτάσουμε λοιπόν. Εμείς προτείνουμε τήρηση του κειμένου της συνθήκης. Αλλά πάντως έχουμε προβλέψει τροπολογίες και για τα δύο. Και εάν παραμείνουμε μέσα στα πλαίσια της συνθήκης, αλλά και αν προχωρήσουμε περισσότερο. Η ανάθεση σε, σε ποιο βαθμό γίνεται, σύμφωνα με ποιο άρθρο, εδώ προ, προτείνεται το 299 άρθρο, αλλά δεν, εδώ δεν δίνει γενική εξουσιοδότηση, άρα πρέπει να εμφανίζονται συγκεκριμένα άρθρα στο κείμενο της Επιτροπής. Αυτό που δεν κάνουμε, και αυτό είναι η πρώτη δική μας παραβίαση της συνθήκης, δεν βάζουμε δηλαδή συγκεκριμένους στόχους, γιατί είναι πάρα πολλοί. Εάν κάνουμε και αυτό, αν πρόκειται να κάνουμε και αυτό, θα το κάνουμε. Έχουμε 30-40 άρθρα όπου η Κομισιόν θέλει να μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές διατάξεις, αλλά δεν βάζουμε εμείς τα όρια μέχρι που μπορεί να φτάσει η Επιτροπή. Εδώ ευχαρίστω να ακούσω δικές σας υποδείξεις. Από την λίστα της Κομισιόν δεν δεχθήκαμε περίπου 12 άρθρα, διότι έχουμε βάλει ήδη τις ε, εκτελεστικές διατάξεις στο ίδιο το νομοθέτημα. Αυτό για την ανάθεση που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω δικαιωμάτων εφαρμογής, ε, συγκρούσεις συμφερόντων, εκτελεστικούς οργανισμούς τα όρια της ανάθεσης των ε, εφαρμοστικών δικαιωμάτων καθώς επίσης και δημοσιονομικούς μηχανισμούς. Πρέπει να συζητήσουμε ακόμη κατά πόσον και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να προβαίνει στην ανάθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρθρο 202. Εδώ δεν θα δοθεί απεριόριστη εξουσιοδότηση από εμά, αλλά θα γίνει προσαρμογή των δύο νομοθετημάτων και έχουμε μάλιστα συντάξει και σχετική τροπολογία. Επίσης, άρθρο 203, ανάκληση της ανάθεσης μετά από πρόταση της ε, Γραμματείας της Επιτροπής να μπορεί δηλαδή να ανακληθεί και κατά τμήματα μόνο η ανάθεση. Δηλαδή να μην αναφερθούμε στο όλον, αλλά μόνο σε τμήματα. Τότε η ανάκληση γίνεται ευκολότερη. Τώρα για την έκδοση της ε, κατανάθεσης νομοθεσίας έχουμε πάλι εδώ περιλάβει την διατύπωση που περιέχει η συνθήκη. Αποδοχή λοιπόν η ένσταση Εδώ αναφερόμαστε πάλι στη συνθήκη. Ο Σάιερ προτείνει αποδοχή η συνθήκη, λέει μονάχα, μονάχα ένσταση. Εδώ είναι ένα σημείο που θα μπορούσαμε να υπερβούμε τα όρια της συνθήκης. Αυτά ήθελα να πω για τις κατανάθεσεις πράξεις. Κάθε φορά υπάρχει και ένα άλλο κέντρο βάρους. Σήμερα το κέντρο βάρους ήταν η κατανάθεση πράξεις. Την επόμενη φορά θα εξηγήσω τα, ολόκληρο το κείμενο της εκθέσεως και για το shared management δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε αγαπητή μας κυρία εισηγήτρια. Διαπιστώνουμε πόσο περίπλοκο είναι ειδικά αυτό το κεφάλαιο. Ο Γκέραν Φέρμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαι επικεφαλής <laughs> δυστυχώς μιας πολύ ολιγομελούς ομάδας σήμερα. Ελπίζω να μην είναι πολύ δύσκολε οι ψηφοφορίε γιατί η σοσιαλιστική ομάδα βρίσκεται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Εγώ ε, ήρθα χθε το απόγευμα, η Φραντσέσκα δεν μπόρεσε να πάει, δεν είναι ότι μποϊκοτάρουμε οι σοσιαλιστές στην Επιτροπή Προπολογισμών. Δεν πρόκειται να επισέλθω σε λεπτομέρειες τώρα στο θέμα τη ούτω ή άλλω οι αρμόδιοι σοσιαλιστές για το θέμα αυτό που σιάζουν σήμερα. Θα επανέλθουμε με πολύ περισσότερα σχόλια στη συζήτηση. Μία γενική τώρα σκέψη για αυτά που είπαμε. Ποια είναι τα προνόμια και εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και φυσικά θα πρέπει να υπερασπιστούμε τις εξουσίες και τα δικαιώματά μας και τα προνόμια μας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το Κοινοβούλιο είναι ένα πολιτικό όργανο και τα προνόμια μας είναι κυρίως πολιτικού χαρακτήρα. Δεν είμαστε ούτε διοικητικό ούτε εκτελεστικό σώμα. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Γιατί αν επισέλθουμε υπερβολικά στις λεπτομέρειες, τότε η εφαρμογή των πολιτικών θα είναι ακόμη, ακόμη πιο δύσκολη. Όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Γιατί θα ε, υπερφορτωθούμε με, με, με μεταφορές, λεπτομέρειες. Ε, δεν θα, χρειαζό, δεν θα μας αρκούν κάποια τρεις βοηθοί. Θα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερους βοηθούς και προσωπικό. Δεν θα πρέπει να επισέλθουμε σε θέματα μικροδιαχείρισης και να αποσπαστεί η προσοχή μας από τα πραγματικά πολιτικά ζητήματα. Θα πρέπει να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα, την ελαστικότητα, να αποφύγουμε την κολυσιεργία της περίτες καθυστερήσει, την ανελαστικότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και φυσικά είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία εδώ. Γιατί αν επικεντρωθούμε μόνο στα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επισέλθουμε σε κάθε λεπτομέρεια, στην παραμικρή λεπτομέρεια σε κάθε θέμα, τότε θα χάσουμε τα πιο βασικά ζητήματα. Θα αποσπαστεί η προσοχή μα Προσοχή για να βρεθεί σωστή ισορροπία. Δεν είναι μόνο τα προνόμια το σημαντικό. Είναι και ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω θεσμικού, πολιτικού θεσμικού οργάνου και θα πρέπει γι' αυτό να βρούμε ένα αποτελεσματικό σύστημα τη εφαρμογή των πολιτικών και κάτι τέτοιο απαιτεί και μια ελαστικότητα. Ευχαριστώ κύριο Σάγκλουντ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ παρόλο που η δική μου ομάδα δεν βρίσκεται στην Αθήνα σήμερα και εμείς δεν είμαστε πολύ στη συνεδρίαση. Για πολλούς και διάφορους λόγους, άνοιξη και λοιπά Είχαμε μία συνεννόηση με το σκιώδη μας παρόντα στη συνομιλία, στις συνομιλίες με την Ίγκε και όπως είπε και ο Γκέραν και ο δικός μας σκιώδης συγητής ε, αυτή τη θέση υποστήριξε. Θα πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία δηλαδή μεταξύ της πολιτικής ευθύνης και της μικροδιαχείρισης. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε την ισορροπία αυτή. Αλλά δεν θα πρέπει να χαθούμε στις λεπτομέρειες. Γιατί έτσι θα διαταραχθεί αυτή η ισορροπία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητά άλλο το λόγο. Δύο παρατηρήσεις. Θα ήθελα από τη μια πλευρά να υπογραμμίσω τα όσα είπατε. Έγκλοντι και Γόραν. Όντως πρέπει να φροντίσουμε ώστε το Κοινοβούλιο να παραμείνει εντός του πολιτικού του ρόλου και να μην αναμεθεί στη διαχείριση. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να βρούμε σωστή ισορροπία με αυτή τη νέα υπόθεση των ε, καταξουσιοδότηση πράξεων. Έχουμε ένα παράδειγμα όταν ε, το Κοινοβούλιο θέλει να παρέμβει στην ε, διαχείριση, είτε πρόκειται για την εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης με διαδικασίες που θα ψηφιστούν σήμερα που απαιτούν κάθε φορά διορθωτικό προϋπολογισμό κάθε φορά που κινητοποιείται το Ταμείο Αλληλεγγύης, είτε με διαδικασία που δεν απαιτεί παρά ένα έμβασμα της χρήσης ε, του Ταμείου για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Ε, διαδικασίες οι οποίες είχαν ε, αρχικά προετοιμαστεί για πολύ λίγε περιπτώσει, αλλά από τη στιγμή που πολλαπλασιάζονται αυτέ οι υποθέσει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα μηχανισμό που επιχρεώνει κάθε φορά να φτάσει το θέμα στι ε, κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, να καθυστερεί η λήψη απόφαση και τελικά χωρί να έχει πολιτική προσθέμενη αξία το Κοινοβούλιο για τι περισσότερε περιπτώσει, χρειάζεται να ψηφίσουμε σύμφωνα με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα αυτή η φιλοσοφία που θέλει να απλοποιήσει και να μην αναμειγνύει τους ρόλους θα πρέπει να εμπνέει τις θέσεις μας και για τον ε, δημοσιονομικό κανονισμό. Και κάτι ακόμα που θέλω να πω, το δεύτερο μάλλον που θέλω να πω, είναι ότι για το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε με τους συντονιστές. Ε, εγώ έλαβα μια επιστολή του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Μα ζητά λίγο περισσότερο χρόνο για να υποβάλουν τη δική τους νομοδότηση, γιατί έχουν πολλά να πούνε για το θέμα αυτό, γιατί ξέρουμε ποια είναι η σημασία του και του Ταμείου Συνοχής των Διευθυντικών Ταμείων στη διαχείριση του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δούμε με τους συντονιστές και κυρίως με την ΕΙΝΚΕ πώς θα προσαρμόσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Να προσθέσω ότι σε ένα τόσο λεπτό ζήτημα, όπως είπε και η ΕΙΝΚΕ, δουλεύουμε επί τη βάση των τροπολογιών στα αγγλικά, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι καθώς θα φτάσουμε στη φάση λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας μας να σεβαστούμε τον κώδικα του πολυγλωσίας. Αυτό είναι αυτονόητο. Ίγκε, έχει σχόλια. Ευχαριστώ για όλα τα σχόλια, αγαπητέ Γιώραν και αγαπητέ Χάκλουντ. Ο στόχος μας είναι κοινό. Και εμείς θέλουμε ένα κείμενο χαρακτήρα πολιτικού, αλλά βέβαια ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι έγγραφο το οποίο απευθύνεται στην διοίκηση. Αυτό που ήθελα εγώ είναι να γνωρίζω ποιο δαπανά τα ευρωπαϊκά χρήματα. Έθεσα λοιπόν ιδιαίτερα το θέμα εδώ της ε, υποχρέωσης απόδοσης λογαριασμών, του υπολόγου δηλαδή, και πώς η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να γνωρίζει κάτι όταν μεταφέρει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες σε κάποιους άλλους ε, στην περίπτωση αυτή λειτουργεί κάπως σαν εποπτικό συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε λοιπόν το εποπτικό συμβούλιο είναι εποπτικό συμβούλιο, είναι αρκετά μακριά από την καθημερινή πράξη. Θέλουμε μια ε, εφαρμογή του κανονισμού μέσω ιδιωτικών τραπεζών. Περί αυτού πρόκειται εν τέλει. Γιατί πρόκειται για τα χρήματα των φορολογουμένων. Άρα να τα αναλάβουν τράπεζες δημοσίου δικαίου. Mm. Τέτοια ερωτήματα μας απασχόλησαν. Απλουστεύσαμε τα πράγματα πολύ. Δώσαμε συγκεκριμένες υποδείξεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα πώς θα λυθεί το πρόβλημα του Ταμείου Έρευνας, επίσης το κόστος του προσωπικού. Μπήκαμε λοιπόν σε λεπτομέρειες και είπαμε ότι παίρνουμε τους υπολογισμούς των χωρών μελών. Και εδώ διευκρινίστηκε το θέμα. Αυτοί, αυτοί οι λογαριασμοί, αυτοί οι υπολογισμοί μάλλον πρέπει να σέβονται ορισμένα κριτήρια. Ούτε και στην Κομισιόν συμφωνούν όλοι βέβαια μεταξύ τους. Υπάρχουν και διαφορετικά συμφέροντα των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Πάντως και εγώ θέλω σίγουρα ένα απλούστερο σύστημα. Το κέριο ερώτημα θα είναι πώς θα γνωρίζουμε και έγκαιρα τι συμβαίνει με τα ευρωπαϊκά χρήματα. Πώς επιτυγχάνονται οι στόχοι μας και γι' αυτό βάλαμε μια στάνταρ τροπολογία που λέει ότι η εφαρμογή εξαρτάται πάντοτε από το γεγονός ότι υπάρχει ένα βασικό δίκαιο, ότι δηλαδή οι ειδικευμένε επιτροπές τα εγγράφουν αυτά και στις βασικές τους νομοθετικές διατάξεις, να, ώστε να καταστεί δυνατόν κάτι που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή άμεση καταβολή σε επιχειρήσεις. Αν εδώ δεν βάλουμε μια τροπολογία, τότε θα φτάσουμε σε χρηματοδότηση πραγμάτων που μόνο εκ των υστέρων θα ανακαλύψουμε ότι είναι δυνατόν να γίνουν. Γι' αυτό θέλω και να είμαστε ε, εξασφαλισμένοι ότι, ότι όταν γνωρίζουμε ακριβώ τι γίνεται να μπορούμε να το παρακολουθούμε. Το Συμβούλιο δικαίω παραπονέθηκε ότι πρόκειται για ενλευκό επιταγή. Γιατί με αυτό το δημοσιονομικό κανονισμό δίνουμε ενλευκό επιταγή στην πραγματικότητα. Εφόσον το πράξουμε πρέπει να γνωρίζουμε πώ θα το πράξουμε και ποιου μηχανισμού ασφαλεία θα περιλάβουμε. Υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες για την ε, περίπτωση των προσωρινών δωδεκατημωρίων. Όπως είπα, υπάρχουν τεχνικές λεπτομέρειες που ε, ασφαλώς μας απασχολούν. Προέρχονται ωστόσο από άλλα έγγραφα και τελικώς καταλήγουν και στο δικό μου. Προσπαθήσαμε να περιλάβουμε και το πολιτικό ενδιαφέρον που έχουμε να υπάρξει καλύτερη, μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό είναι προς το δικό μας, αυτό είναι το δικό μας ενδιαφέρον. Μπορούμε να βελτιώσουμε εκεί την κατάσταση και στην κοινή διαχείριση, το shared management, υπάρχει μια νέα συστημική πρόταση, το άρθρο 56 δηλαδή, που ακόμα δεν γνωρίζουμε λεπτομερώς ποιες είναι οι επιπτώσεις της εφαρμογής του, αλλά πάλι εδώ πρέπει να προσέξουμε να μην προκαλέσουμε χάος. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα μαζί σας με την έννοια αυτή. Ορισμένα πράγματα βέβαια ηχούν περίπλοκα, αλλά δεν είναι. Αυτό που ήθελα εγώ είναι να διατηρήσουμε την γνώση του τι γίνεται, που καταλήγουν τα χρήματα των φορολογουμένων. Αυτό το χρωστάμε στους ψηφοφόρους μας. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Οποιουσδήποτε θέλει να με ερωτήσει ανα πάσα στιγμή, ημέρα και νύχτα είμαστε πανέτοιμοι και πανέτοιμες να απαντήσουμε. Μέχρι τώρα κανείς δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον βέβαια να μάθει οτιδήποτε. Και αυτό δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε τόσο πολύ. Ας, ασχοληθούμε με την ουσία του θέματος και όχι με ε, ε, επιχειρήματα που ε, δεν οδηγούν πουθενά. Δεν θέλω να μπούμε σε μικροδιαχείριση, αλλά υπάρχει κίνδυνος όπως πήγαιναν τα πράγματα, όπως άλλωστε προσπαθεί συνήθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπάθησε να μεταθέσει τις ευθύνες για την δαπάνη των χρημάτων, προτιμώ να την αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευθύνη αυτή και αυτός είναι ο στόχος της έκθεσης και των τροπολογιών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ίγκε. Μπορούμε να απελευθερώσουμε την Ίγκε που έχει άλλες υποχρεώσεις. Και να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Κατ' εξαίρεση να κάνουμε τις ψηφοφορίες για τα εμβάσματα για να μπορέσει να αποχωρήσει και η Χέλγα. Helga, έχεις κάποιες ε, μεταφορές. Ευχαριστώ. Ναι, η ομάδα μου πάει στη Βουδαπέστη σήμερα. Γι' αυτό και πρέπει να αποχωρήσω εντός ολίγου. Λοιπόν, έχει ζητηθεί μεταφορά, μεταφορά που αφορά τις τροποποιήσεις στο πρόγραμμα θέσπισης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών. Η τροποποίηση στο σχέδιο εγκατάστασης της ΟΚΕ θα οδηγήσει σε δημοσιονομικές εξοικονομήσεις και θα ήθελα να σας ζητήσω κύριε Πρόεδρε να βάλετε σε ψηφοφορία αυτήν τη μεταφορά και συστήνω να την εγκρίνετε. Ευχαριστώ. Τα δύο ταυτόχρονα. Ε, ε, ε, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Ξέρετε από τους συναδέλφους. Donc, nous a présenté Ωραία. Η Έλγα μας παρουσίασε αυτά τα δύο αιτήματα που είναι αρκετά απλά. Θα ψηφίζουμε από κοινού ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δύο κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Εγκρίνονται λοιπόν. Ευχαριστώ Χέλγα. Μπορείς να φύγεις για την Βουδαπέστη. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, Επαναρχόμαστε στην προβλεπόμενη ημερήσια διάταξη, το σημείο 4 προετοιμασία ε, του προπολογισμού για το 2012. Εχθές είχαμε ένα τριμερή διάλογο και θα δώσω το λόγο στη Φραντσέσκα Μπαλτζάνη που με την ευκαιρία αυτού του τριμερούς διαλόγου παρουσίασε τους προσανατολισμούς του Κοινοβουλίου. Φραντσέσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εχθέ έγινε ο τριμερής διάλογος για τις γραμμές του προπολογισμού για το 2012. Ένας πολύ απλός τριμερής διάλογος γιατί σε αυτή τη φάση ακόμα δεν έχουμε αριθμητικά στοιχεία. Οπότε είναι σαφώς πιο εύκολο να μιλάμε για τις προτεραιότητε του προπολογισμού. Εγώ παρουσίασα τις κατευθύνες γραμμέ που ψηφίσαμε. Ιδιαίτερα όσον αφορά την στρατηγική 2020. Προσπάθησα δηλαδή να υπογραμμίσω ότι στο κέντρο του επόμενου μας προϋπολογισμού είναι η στρατηγική 2020, πράγμα που σημαίνει και ένα μέγα αίτημα συνοχής, συνέπειας από πλευράς Κομισιόν και Συμβουλίου, γιατί δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μια στρατηγική για την ανάκαμψη της Ευρώπης μέσω και μακροπρόθεσμα, αν δεν αποφασίσουμε συγκεκριμένα να εργαστούμε από αυτού και με επικοδομητικό πνεύμα. Προσπάθησα επίσης να υπογραμμίσω πως είναι ένας καλός προπολογισμό σε ένας προπολογισμό ε, σε περίοδο κρίσης δεν αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με το πώς θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική παγίωση άσχετα από το περιεχόμενό της ε, με μαθηματικό τρόπο δηλαδή. Αντίθετα πρέπει να υπάρξει ένας προπολογισμό που θα δίνεται μεγάλη προσοχή στο περιεχόμενο. Ένας, μια μαθηματική αύξηση των πληρωμών δεν σημαίνει ότι είναι η σωστή απάντηση σε μια φάση κρίσης γιατί είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε με ακρίβεια που ε, θα αυξηθούν οι πληρωμές και επίσης πού θα αυξηθούν οι υποχρεώσεις, που είναι τα κομμάτια του, που, ποια είναι τα τμήματα του προϋπολογισμού που αφορούν το μέλλον και που θα υποδείξουν σε ποιου τομεί θέλει να επενδύσει η Ένωση. Ζήτησε επίσης να εξεταστεί προσεκτικά το ψήφισμα σε εκείνα τα σημεία όπου ζητάμε να γίνουν μεταφορές carry over τα ποσά τα οποία δεν δαπανήθηκαν πέρυσι, ώστε να έχουμε περισσότερους πόρους και ένα είδος οριζόντιας ευελιξίας στο διαχρονικά η αντίδραση περισσότερο μάλλον το κλίμα που επικράτησε γιατί δεν ήταν δυνατόν να μπούμε σε λεπτομέρειες όπω καταλαβαίνετε ε, το κλίμα ήταν μάλλον θετικό κυρίως όσον αφορά την ανάγκη να επενδύσουμε στην στρατηγική 2020 που επαναλαμβάνω είναι η αληθινή απάντηση πιο χρήσιμη των πολιτικών λιτότητα ε, σε σχέση με την κρίση και η Ουγγρική Προεδρία Μα είπε επίση ε, αρχικά ότι συμφωνεί με την ανάγκη βέβαια να υπάρχει ένας ισχυρό προπολογισμό για το 2012. Σα θυμίζω επιπλέον γιατί αυτή η Επιτροπή είναι πια στο τέλο Μαρτίου ότι θα πρέπει σε αυτή τη φάση να επικεντρώσουμε την προσοχή στα πιλωτικά προγράμματα και τι προπαρασκευαστικέ δράσει. Και το θυμίζω αυτό γιατί ο στόχο είναι ο εξή. να παρουσιάσουμε μέσω ε, μέχρι τον Ιούνιο ένα προσωρινό κατάλογο στην Κομισιόν για να έχουμε μια πρώτη αντίδραση και οργανώνουμε και μια ακρόαση για να κατανοήσουμε ποια πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικέ δράσει δεν λειτουργούν καλά, ποια είναι επιτυχία αντίθετα και άρα να κατανοήσουμε πώς θα προσανατολιστούμε καλύτερα στην προετοιμασία της πρότασης για το 2012 με στόχο να αποφύγουμε καθώς αυτά τα προγράμματα και αυτές οι δράσεις παίρνουν τμήμα του περιθωρίου, δηλαδή περιορίζουν το περιθώριο που είναι ούτως ή άλλως μικρό ε, να δούμε ακριβώς ποιες δράσεις έχουν πιθανότητες επιτυχίας και να μην ε, δεσμεύσουμε άσκοπα χρήματα. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Συμπληρώνοντας αυτά που εξαιρετικά, με εξαιρετικό τρόπο μας εξέθεσε η Φραντζέσκα, θα ήθελα να προσθέσω ότι ο τριμερής διάλογος για την κατάρτιση του προπολογισμού του 2012 και την κατάσταση προβλέψεων για το 2012 δεν ήταν μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων ως ήθιστε σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε στις αρχές του χρόνου αλλά ουσιαστικά ήταν η εκφώνηση δύο μονομερών ομιλιών. Το Συμβούλιο εξήγησε γιατί ζητά τη μέγιστη δημοσιονομική λιτότητα και η Φραντσέσκα παρουσίασε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση τους γενικούς προσανατολισμούς. Το θετικό, όπως μας είπε η Φραντσέσκα, είναι ότι και από τις δύο πλευρές τις τρεις μάλλον μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το βασικό μέλημα είναι να ληφθεί υπόψη και σημαντικό σημείο αναφοράς η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το 2020. Και έτσι θα διευκολυνθεί η συμφωνία για τις προτεραιότητες. Αυτό που είναι κάπως απογοητευτικό είναι ότι οι συνομιλητές μας ε, σε στον τριμερή διάλογο και ιδιαίτερα η Ουγγρική Προεδρία είναι δεμένη χειροπόδαρα από τις προηγούμενες αποφάσεις ε, σε επίπεδο ε, γραμματεία συμβουλίου και μόνιμης αντιπροσωπείας. Και το λέω αυτό παρουσία των εκπροσώπων της Ουγγρικής Προεδρίας. Είναι δεμένη χειροπόδαρα. Ακούμε μόνο ξύλινη γλώσσα. Θα μπορούσαμε να μην έχουμε καν τριμερή διάλογο και να πώ έχουμε μια ανταλλαγή εγγράφων. Και με ε, και έμεινα εμβρόντιτος γιατί δεν έγινε κανένα σχόλιο. Τελείως no comment. Και παρά την μεγάλη ικανότητα πυθού, την τεράστια ικανότητα πυθού που διαθέτω και που έφτασε στα ωριά τη. παρόλο που στο πλαίσιο που βρεθήκαμε Όπως είχα κάνει και στην ιδιωτική συνομιλία με τους ενδιαφερομένους πριν από μερικές εβδομάδες, επανέλαβα την έκκλησή μου για να επανέλθουμε σε μια πρακτική που εφαρμόζαμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια και την εγκαταλείψαμε για άγνωστους για μένα λόγους. Συγκεντρώνουμε την πολιτική συζήτηση στα νούμερα ε, μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά τις ε, πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων και όχι τις πιστώσεις πληρωμών. Όπως μας υπενθύμησε ο Γκόραν, είμαστε πολιτικά όργανα. Και τα πολιτικά όργανα ενδιαφέρονται για τις αναλήψεις υποχρεώσεων, για τις πολιτικές επιλογές ε, που μεταφράζονται σε αναλήψη υποχρεώσεων. Από τη στιγμή που έχουν αναλυφθεί υποχρεώσεις θα πρέπει να καταβληθούν και οι πληρωμές. Οι πληρωμές είναι οι μαθηματικές, νομικές, αναπόδραστες συνέπειες των ηλυμένων υποχρεώσεων. Και όπως κάθε συζήτηση, και πέρυσι για παράδειγμα που συζητήσαμε το προϋπολογισμό το 2011, στη συζήτηση μονοπόλησαν οι πληρωμές, μας οδήγησαν φέτος σε ένα διέξοδο. Γιατί τα τελευταία χρόνια μόνο στι πληρωμές είχαμε επικεντρωθεί. Και μετά από προηγούμενες αποφάσεις και μετά από την αύξηση του καθεστώτος των ε, διαρθρωτικών ταμείων και τις προσπάθειες αύξησης των δαπανών με το πρόγραμμα ανάκαμψης προκειμένου να στηρίξουμε την οικονομία εν μέσω της κρίσης. Τώρα θα αυξηθούν οι πληρωμές για πρώτη φορά το 2011 και μετά το 2012. Αν συνεχίσουμε λοιπόν να περιοριζόμαστε στο να λέμε ότι θέλουμε δημοσιονομική λιτότητα και στις 27 χώρες, 27 κρατικούς προϋπολογισμούς και στον κοινοτικό και να επικεντρώνουμε την πολιτική συζήτηση πληρωμές, τότε θα οδηγηθούμε σε διέξοδο και σε παράδοξο. Αυτό υποστήριξα και στον τριμερή διάλογο και το δηλώνω εδώ και δημοσίω γιατί μας ακούει και ο κόσμος. Θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου αλλά και την απογοήτευσή μου. Γιατί δυστυχώς αυτή μου η έκκληση δεν προκάλεσε καμία αντίδραση. Ούτε θετική, ούτε αρνητική. Άφησε τους πάντες αδιάφορους και προσέκρουσε σε ένα ε, αυτισμό, σε μία σιωπή εκ μέρους των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων. Αυτό θα ήθελα να σας ενημερώσω. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Έχοντας υπόψη ότι σε λίγο θα κληθούμε να λάβουμε μία απόφαση για τις πιστώσεις πληρωμών του 2011. Και εκεί θα γίνουμε μάρτυρες αυτής της πολιτικής αντίφασης που βιώνουμε σήμερα, και που δεν θα είναι η μόνη δυστυχώς. Και με βάση όλες τις ενδείξεις που έχουμε και τις υποδείξεις που μας έκανε ο, κύριος, ο Επίτροπος και όταν ήρθε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και από πληροφορίες που είχαμε για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012 γνωρίζουμε ότι για νομικούς λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποχρεωθεί να μας προτείνει αύξηση των πιστώσεων πληρωμών που θα φαίνεται ότι αυξάνονται κατά μεγάλο ποσοστό, ενώ στην ουσία είναι η εκτέλεση των προηγουμένων αποφάσεων, των πολιτικών αποφάσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων. Άρχεται η συζήτηση. Ο κύριος Μπόκρος. Ευχαριστώ. Μία σύντομη παρατήρηση καταρχήν. Θα ήθελα εδώ στην συνεδρία τη Επιτροπή Προπολογισμών, θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη μου απογοήτευση για το γεγονό ότι οι συντονιστές των μικρών ομάδων αποκλείστηκαν από το χθεσινό τριμερή διάλογο. Πώς είναι δυνατόν να εκτελέσουμε τα καθήκοντα που έχουμε απέναντι στι ομάδες μας, να τους ενημερώσουμε, και να τους τροφοδοτήσουμε με έγκυρες πληροφορίες εφόσον μας αποκλείεται από σημαντικές συνεδριάσεις όπως ήταν αυτή του τριμερούς διαλόγου. Ελπίζω είναι η τελευταία φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο με τέτοια περιθωριοποίηση των συντονιστών των μικρών ομάδων. Ευχαριστώ αγαπητή συνάδελφα. Ο Σελβαντόρ Γκαρίγκα. Ευχαριστώ. Ο συντονιστής του ΕΛΚ θα ήθελα να εκφράσω την ε, συμφωνία μου και την υποστήριξή μου προς τον πρόεδρό μας, τον Αλένα Μασούρ. Πέραν της απόφασης που θα κληθούμε να λάβουμε για τις πιστώσεις πληρωμών του 2011. Θα ήθελα εδώ να αποτανθώ στην εισηγήτρια του προϋπολογισμού του 2012, την κυρία Μπαλτσάνη, και να πω ότι η κατάσταση πραγματικά θα είναι δύσκολη και είχαμε μια πρόγευση στον χθεσινό τριμερή διάλογο για το πόσο δύσκολη θα είναι η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη κατανάλωση των πιστώσεων πληρωμών το 2012 και 2013, μεγαλύτερη από ό,τι το 2011. Και το 2011 η αναλήψη υποχρεώσεων που έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο ήταν απολύτως ανεπαρκής για να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες των πολιετών μας συμφωνιών για τα διαρθρωτικά ταμεία για παράδειγμα αλλά και για άλλα θέματα όπως είναι η εφαρμογή του Ταμείου Ελεγγύης που προϋποθέτουν πολύ πιο πενιχρά Αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε καταρχήν, ε, κυρία Βαλτσάνη, είναι να αποφύγουμε να, να φτάσουμε τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο ε, μπροστά σε μια νέα μονομερή διακήρυξη του Συμβουλίου που θα επιβάλλει μονόπλευρα μία μείωση των πιστώσεων πληρωμών σε ένα επίπεδο που θα καθιστά δύνατη οποιαδήποτε εκτέλεση του προϋπολογισμού. Βέβαια, η διοργανική διακήρυξη για να εξασφαλιστεί η εκταμείευση συμπληρωματικών δαπανών δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο και αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη η συγκεκριμένη στη στρατηγική τη. Εμεί θα τη στηρίξουμε στο θέμα αυτό, γιατί είναι το πιο σοβαρό ζήτημα κατά τη γνώμη μα. Είναι αδύνατο να έχουμε ένα κοινοτικό προπολογισμό με ανεπαρκείς πιστώσεις πληρωμών, με πιστώσει πληρωμών που δεν μα επιτρέπουν να, να ε, ικανοποιήσουμε τι στοιχειώδεις μα ανάγκε. Και κάτι που υπενθύμησε ο Επίτροπο Λεβαντό και στον τριμερή διάλογο είναι τι θα γίνει με το πρόγραμμα ITER του, πυρηνικού θερμο, του θερμοπυρηνικού πειραματικού αντιδραστήρα. Ήταν σαφές ότι οι πιστώσει του 2010 χάθηκαν, οπότε οποιαδήποτε απόφαση για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ITER θα πρέπει να προέλθει από τον προϋπολογισμό του 2012. Κάτι που θα είναι πολύ δύσκολο ε, να βρεθεί ένα τέτοιο κονδύλιο, συμπληρωματικά δηλαδή κονδύλια και πιστώσεις για το πρόγραμμα ITER. Πάντως υπάρχει ε, η υποχρέωση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η δέσμευση που έχει αναλάβει και που λύγει το 2012. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν ή συμπληρωματικέ πιστώσει, δεν ξέρω από εκεί που δεν υπάρχουν, ή να βρούμε κάποια κονδύλια για να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας για το ίτερ. Δύσκολο λοιπόν θα είναι το έργο τη εισηγήτρια. Αλλά σε ό,τι αφορά τι πιστώσει πληρωμών, νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε όλε οι ομάδε και να ακολουθήσουμε μια κοινή στρατηγική. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Η Χέλγα που είναι ακόμα εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια παρατηρήση ότι συμμερίζομαι τις ανησυχίες του κ. Μποκρός ότι δηλαδή είναι η καλύτερη διαδικασία να αποκλείονται οι συντονιστές των μικρών ομάδων από αυτούς τους τριμερείς διαλόγους. Α, τώρα, Πρόεδρε, με την πρότασή σας ε, να εστιαστούμε στο θέμα των υποχρεώσεων. Πολύ καλή, ευφυής και σημαντική ιδέα. Α, και λυπάμαι που το Συμβούλιο ε, δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε σε αυτό. Αυτό βέβαια κατοπτρίζει το πολιτικό πρόβλημα που έχουμε ε, να αντιμετωπίσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά η Κομισιόν το συνειδητοποιεί πως φυσικά με τις, υποχρεω... με τις πληρωμές λόγω υποχρεώσεων που έχουμε είναι απαραίτητο να εστιάσουμε την προσοχή στο θέμα των πιστώσεων ε, των υποχρεώσεων για το θέμα του Ταμείου Αλληλεγγύης. Νομίζω πως Πρέπει να επιμείνουμε για το θέμα της δήλωσης περιπιστώσεων και να μιλήσω για το ίτερ. Να ξέρω πως δεν σας εντυπωσιάσει πως εμείς οι πράσινοι είμαστε κατά τέτοιου είδους επενδύσεων γιατί θεωρούμε πως είναι επικίνδυνη η τεχνολογία και ότι πραγματικά θα πρέπει να γίνουν τεστ αντοχής εκεί και θα πρέπει να υπάρχουν τρόποι ε, για να ε, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πρώτα, πριν να φτάσουμε στην σύνδεξη. Ξέρω πως ε, στη χώρα μου και στη Γαλλία είναι πολύ αναπτυγμένη η πυρηνική ενέργεια, αλλά πρέπει πλέον ως Ευρωπαίοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της πυρηνικής ενέργειας και δεν πρέπει μόνο να ακολουθούμε τη γραμμή της Κομισιόν και να βρούμε τα χρήματα στον προπολογισμό του 2012, αλλά να έχουμε μια γενικότερη προσέγγιση στα προβλήματα αυτών των τεχνολογιών. Ευχαριστώ. Euh, euh, Ευχαριστώ, Χέλγα, για το σχόλιο σου. απαντήσω, γιατί ίσως και άλλοι θα κάνουν τις ίδιες παρατηρήσεις, για τη σύσταση της αντιπροσωπείας στους τριμερείς διαλόγους. Εγώ κάπως εντυπωσιάζομαι από τα σχόλιά σας δεν κάνουμε παρά να εφαρμόσουμε την ομόφωνη απόφαση των συντονιστών. Λήφθη αυτή στις 10 Φεβρουαρίου 2010 και μάλιστα είναι παράδοση στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών και εκείνη την ημέρα αποφασίσαμε για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιπροσωπεύεται η Επιτροπή Προϋπολογισμών σε όλες τις εξωτερικές εκδηλώσεις. Τριμερής διάλογος, αλλά επίσης κατανομή για τις μελέτες, για τις ακροάσεις, ε, για τις διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και με την ε, Επιτροπή του Συμβουλίου για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και κοινή ε, ασφάλειας, την ομάδα εργασία, την αποστολή αντιπροσωπείων, Και όσον αφορά τους τριμερείς διαλόγους αποφασίσαμε σύμφωνα με μια αρχαία πρακτική, παλιά πρακτική, ότι η αντιπροσωπεία θα περιορίζεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και τους εισηγητές για τα θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη. Και τελεία και παύλα. Με δυνατότητα για κάθε ομάδα που το επιθυμεί να έχει έναν εκπρόσωπο στο επίπεδο των βουλευτών υπαλλήλων και των βοηθών. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως στον τριμερή διάλογο δεν μπορεί να υπάρχει παρά μόνο ένας εκπρόσωπος και μόνο ένας να μπορεί να λάβει το λόγο στο όνομα του Κοινοβουλίου και απέναντί μας με τον ίδιο τρόπο έχουμε μόνο έναν πολιτικό που είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και ο Επίτροπος. Τελεία. Και την περασμένη χρονιά φρόντισα και θα συνεχίσω να φροντίζω ούτως ώστε κάθε φορά που θα έχουμε πραγματικά έναν τριμερή διάλογο με πολιτικό χαρακτήρα να βρίσκεται γύρω από το τραπέζι, να βρίσκονται γύρω από το τραπέζι και άλλοι πολιτικοί εκπρόσωποι ανάλογα με το θέμα. Γιατί όπως είπε και ο κ. Ποκρός, βέβαια θα είναι εκεί αλλά θα είναι βουβή. Όλοι μπορέσαν να εκφραστούν, ε? και το αποφασίσαμε στην προσυνδιαλλαγή που όπως την είπαμε με το Προεδρείο του ε, Κοινοβουλίου για να συνδυάσουμε και να μιλήσουμε για τις εκτιμήσεις για το 2012. Νομίζω πως με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε. Κύριε Αγγλούντ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. σημειώνω αυτό που είπατε καθώς και την υπόσχεση που δώσατε χθε. και τα εκτιμώ εμείς της ομάδας των φιλελευθέρων εκτιμούμε το ότι υποσχεθήκατε ότι στο μέλλον σε τριμερείς διαλόγους με κάποια σημασία θα εκπροσωπούνται οι ε, πολιτικές ομάδες Τουλάχιστον είχαμε πει στις 10 Φεβρουαρίου ότι θα, στις 2 Φεβρουαρίου μάλλον, στη συμφωνία που αναφέρατε, ότι θα <clears throat> εκπροσωπούνται τουλάχιστον με ε, μέλη της γραμματείας. Βέβαια, όταν είναι 20 εκεί θα μιλούμε μέσω του ε, εισηγητού. Αλλά μπορούν θαυμάσια να είναι παρόντες και οι συντονιστές, έστω και αν δεν λαμβάνουν το λόγο. Και οι ε, πολιτικοί μας σύμβολοι οι οποίοι μας μεταφέρουν και τις πληροφορίες. Είναι ζήτημα προσέγγισης. Και αυτό ίσως θα πρέπει να ξανασυζητηθεί κάποια στιγμή στους συντονιστές γιατί φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα πλέον για τις μικρές ε, πολιτικές ομάδες. Πάντως, όπως είπα, ε, δεχόμαστε την υπόσχεση που έδωσε ο Πρόεδρος εχθές και μας ικανοποιεί. Σας ευχαριστώ αγαπητέ ε, συνάδελφε. Ο κύριος Φάρμ. Για τον τριμερή διάλογο πρώτα. Δεν θα μπω περισσότερο στο θέμα αυτό, αλλά πρέπει να σκεφτούμε λίγο και την ροή των πληροφοριών. Βέβαια δεν μπορούν να είναι όλοι παρόντες, διότι θα, θα ξεπέρναγε τα όρια πλέον ε, ποσοτικά. Αλλά πρέπει να μεταφέρονται οι πληροφορίες. Τώρα, για τις υποχρώσεις και τις πληρωμές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σύμφωνο με την Χέλκα και ε, με άλλους συναδέλφους που είπαν ότι οι προτεραιότητές μας είναι φιλόδοξε στι υποχρώσεις, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα. Όπως είδαμε και πέρσι το Συμβούλιο, δέχθηκαν αρκετά γενναιόδωρα ε, τις υποχρεώσεις, αλλά ήταν απόλυτα άκαμπτοι ε, στις ε, πληρωμές. Δεν ξεπέρασαν με κανένα τρόπο το ποσοστό που προβλεπόταν. Και αυτό σημαίνει ότι αρχίζει και μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ υποχρώσεων και πληρωμών. Και το Συμβούλιο φαίνεται ότι θέλει να κόψει τον ομφάλιο λόγο μεταξύ υποχρώσεων και πληρωμών. Όπου μπορεί να φτάσουμε σε μια κατάσταση που θα απορρίπτουν πληρωμέ, που ε, θα ρίχνουν το βάρο στην μη εφαρμογή πολιτικών, ώστε να εξευρεθούν πόροι για μια αναδιάρθρωση για να μπορούν να πληρώνουν τις δικές τους προτεραιότητες και τότε θα φτάσουμε σε ε, ένα πολιτικό χάο. Πρέπει να το σκεφτούμε περισσότερο όχι να πούμε ότι οι υποχρεώσει είναι οι προτεραιότητε μα. Τι θα πει η υποχρέωση εάν αυτή δεν πρόκειται ποτέ να εφαρμοστεί. Ε, πρόκειται για αέρα κοπανιστό. Άρα πρέπει να μην κοπεί ο σύνδεσμο αυτό μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών και πρέπει να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος σε αυτόν τον σύνδεσμο. Όχι να πούμε μάλιστα φιλόδοξη υποχρεώσει και μετά δεν ε, μας ενδιαφέρει ε, τίποτε περισσότερο. Εν τέλει για το ΙΤΡΕ, για το ΙΤΕΡ μάλλον συγγνώμη είναι απογοητευτικό. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που πάει να γίνει ε, νομική μάχη. Θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για το 2010. Το 2010 ακόμα νομίζουμε πως όχι. Οι νομικές υπηρεσίες του Συμβουλίου λένε όχι. Άρα δεν μπορούμε. Για μας ένα πράγμα είναι σαφές. Δεν μας ενδιαφέρει εάν μπορούμε να βρούμε από το 2010 ή το 2011 κάποιο περιθώριο που δεν εξαντλήθηκε ή νέα χρήματα για το 2012 αλλά δεν δεχόμαστε ε, να ληφθούν χρήματα από άλλες προτεραιότητες υπέρ του ΙΤΕΡ από το πρόγραμμα ε, έρευνας, από το πρόγραμμα έρευνας. Μιλούμε για 500 περίπου ε, εκατομμύρια ευρώ. Να φύγουν αυτά από άλλες γραμμές του προπολισμού του Ταμείου Έρευνας για να πάνε στο ΙΤΡΕ. δεν έχει ακόμα λυθεί το πρόβλημα του redeployment και για μας είναι πάρα πολύ επίμαχο. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Εδώ έχω δύο σχόλια για τις πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών. Ίσως εδώ πρέπει να τεθεί υπό την ισχύ του δημοσιονομικού κανονισμού, γιατί οι πιστώσεις πληρωμών είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικές δαπάνες. Έχουμε καταργήσει βέβαια την διάκριση αυτού που λεγόταν τότε και κακός ε, πιστός, υποχρεωτικές ή μη υποχρεωτικέ πιστώσεις. Αλλά στην ουσία αυτό είναι. Και ο Γιώραν έχει δίκιο που λέει ότι εάν επιμείνουμε ώστε να επικεντρωθεί η συζήτηση στις πιστώσεις υποχρώσεων, δεν έχει άλλο νόημα αυτό παρά μόνο εάν οι πιστώσει πληρωμών θεωρηθούν πλέον πιστώσει υποχρεωτικέ. Αν από την άλλη μεριά το Συμβούλιο βρήκε τον τρόπο να διακρίνει, να απομακρύνει τις δύο αυτές κατηγορίες, τότε μπαίνουμε σε μια επικίνδυνη κατάσταση, κατάσταση εντελώς σουρεαλιστική. Και ασφαλώς ε, πρέπει ο, ο εισηγητής μας να εγγύψει το θέμα αυτό. Για το ΙΤΕΡ έχει λήξει η διαπραγμάτευση για το 2010, για τον προπολογισμό 2010. Μένει να δούμε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κάτι και τι για τον προπολογισμό του 2012. Οπότε μπορούν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, όπως άλλωστε το είπε και ο ίδιος αναφερόμενος και στην, ε, θέση της ομάδας. Λάσλο Σούριαν. Λάσλο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα κύριε Πρόεδρε, λίγα λόγια για το ίδιο, το, για το ίδιο αυτό θέμα. Εάν το Συμβούλιο στην διάρκεια των διαπραγματεύσεων του προϋπολογισμού εξετάζει τις πιστώσεις πληρωμών και κάνει προτάσεις για υπερβολική περικοπή τους, τότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Έχετε όλη η μετάφραση. Μου φαίνεται πως τα γαλλικά δεν λειτουργούν. Δεν, δεν ακούω μετάφραση στα γαλλικά. Τα γαλλικά λοιπόν ακούγονται τώρα. Έχει καλώ. Τώρα σα ακούω. Λάσουλα, έχετε πάλι το λόγο. Αρχίζω από την αρχή, ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, εάν το Συμβούλιο επιθυμεί να μειώσει, να περικόψει δραστικά τις πιστώσεις ε, πληρωμών, εμείς θα πρέπει να τις υπερασπιστούμε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του προϋπολογισμού, εφόσον θεωρούμε ότι μειώνονται υπερβολικά οι πιστώσεις όπως έγινε πέρσι. Η συζήτηση στρέφεται κατά πρώτο λόγο όχι γύρω από τις ε, μακροπρόθεσμες υποχρώσεις και γι' αυτό ε, ε, αναγκαστήκαμε να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος στις ε, πιστώσεις πληρωμών. Είναι ενδιαφέρον να δούμε στο ετήσιο σχέδιο του προϋπολογισμού όταν θα κάνουμε το σχέδιο αυτό οι συζητήσεις στρέφονται κυρίως γύρω από τις πιστώσεις πληρωμών και ένα μικρό μέρος εξετάζει τις ίδιες τις πληρωμές. Ίσως αυτό να είναι ορθό, αλλά εάν κανείς κάνει τον κόπο να προσθέσει τις ε, πιστώσεις των υποχρώσεων στο επταετές πρόγραμμα θα δει ότι το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από τις πληρωμές. Είναι δηλαδή ήδη προκαθορισμένη αυτή η ένταση. Ε, είναι ενταγμένη η ένταση αυτή μέσα στο σύστημα και κάθε χρόνο όταν έχετε μια χώρα μέλος και θέλει και ζητεί πιστώσεις πλωμών και φτάνουμε πλέον στην οροφή αναγκαζόμαστε να λειτουργούμε σαν πυροσβεστική υπηρεσία δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε χρήματα στη βάση μεταφορών πιστώσεων έχουμε λοιπόν εδώ δύο επίπεδα της συζητήσεως και αυτά πρέπει κάπου να εξισορροπήσουν και αυτό και για την επόμενη επταετή δημοσιονομική προοπτική. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να επανέλθει. Είπε ο Πρόεδρος ότι εξεπλάγει από το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν αντέδρασε στην πολύ λογική πρόταση που έγινε. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε ακριβώς. όσον αφορά τα ποσά. αλλά βλέποντας προς το μέλλον, εάν θέλουν οι χώρες μέλη να χρησιμοποιήσουν και τα υπόλοιπα, έχουμε ωστόσο κάποιους περιορισμούς μέσα στους οποίους οφείλουμε να χειριστούμε τον προϋπολογισμό. Οι χώρες μέλη μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Βέβαια μέχρι τώρα ποτέ δεν έγινε κάτι τέτοιο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα εξομάλυνε ή τέλος πάντων διέσωσε την κατάσταση λειτουργώντας ως πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Το Συμβούλιο δεν είχε την ευκαιρία καν να απαντήσει μέχρι τώρα, διότι οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου δεν εκπροσωπούσαν ούτε καν τις χώρες τους, αλλά τις 27 χώρες μέλη. Και δεν είχαν εντολή να πούν οτιδήποτε για ένα θέμα τέτοια σημασίας και με τόσο σημαντικέ επιπτώσει για το μέλλον. Στην ουσία λοιπόν οι συγγύοι που τήρησαν την απάντησή τους. Ο κ. Μπόκρος ωστόσο έχει λάθος όταν μιλεί για, το, για τη σύνθεση των ε, συντονιστών που λέει ότι αποκλείστηκαν οι συντονιστές των μικρών πολιτικών ομάδων. Όλοι οι συντονιστές αποκλείστηκαν. Είχαμε βέβαια παρόντα τον Σαλβαδόρ Γαρίγα, αλλά όχι υπό την ιδιότητά του συντονιστού. Ήταν διότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει ο εισηγητής μας. Και ο συντονιστής των σοσιαλιστών αποκλείστηκε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, αποκλείστηκε. Όλοι οι συντονιστές λοιπόν έμειναν εκτός. Η Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο επίσης αποκλείστηκαν από την πλευρά του Συμβουλίου. Πρόκειται για μια πρακτική την οποία είχαμε και στο παρελθόν και βρίσκω ότι είναι ορθή. Μιλούμε για ένα σχετικά περιορισμένο ε, σε σημασία τριμερή διάλογο και επομένως σημασία έχει να παρευρίσκονται οι εισηγητές των οποίων τα θέματα συζητούνται. Νομίζω ότι χάρη στη γενεοδορία του Προέδρου όταν μιλήσαμε όταν μιλούμε μάλλον για σημαντικά θέματα, ήταν διατεθειμένος να επιτρέψει και σε ορισμένους συντονιστές να συμμετάσχουν στην ομάδα αυτή. Όμως όπως ακούσαμε πρόκειται για παρουσία σιγή διότι το κοινοβουλίο μιλεί με μια φωνή και όχι με τρεις ή τέσσερις, γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε σε θέση να ε, προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας απέναντι στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δε πολιτικές ομάδες το δέχθηκαν αυτό μέχρι τώρα. Το ότι θα πρέπει να παρίστανται οι δικοί μας εμπειρογνώμονες, αυτό πάντοτε είναι δεκτό. Βέβαια η γραμματεία συντάσσει σύνοψη των συζητήσεων και την διαβιβάζει. Ε, καμιά φορά βέβαια εκεί μεταφέρονται και υποκειμενικές απόψεις. Όταν μιλούμε για εμπειρογνωμοσύνη, θα πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια να μεταφέρονται οι απόψεις μας. Όπως είπα, ήταν η γενναιόδορη στάση του Πρόεδρου και εγώ την υποστηρίζω. Αρκεί να μην σημαίνει ότι αυτό θα θεωρηθεί αργότερα προηγούμενο και τελικώς θα καταλήξουμε με μια αντιπροσωπεία οκταμελή ή εννιαμελή που θα πηγαίνει εκεί κάθε φορά. Η γενεοδορία του Προέδρου δεν δημιούργησε προηγούμενο. Ο κύριος Χάρτονγκ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση ως προς την έκβαση του τριμερούς διαλόγου. Για την ανάληψη υποχρεώσεων τώρα, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι συνέβη πέρυσι. Οι αρχές οφείλουν να είναι υπεύθυνε και αξιόπιστες. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα εξοικονόμηση στον προπολογισμό. Ο Επίτροπο Λεβαντόφσκι πραγματοποίησε επίσκεψη την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή τη Ολλανδία και μίλησε για την θέσπιση ενό ευρωπαϊκού φόρου για να δημιουργηθούν περισσότερα κοινοτικά έσοδα αντί να περικοπούν οι δαπάνες και νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο αντί να προσθέτουμε νέους φόρους να είμαστε πιο ορθολογικοί στις δαπάνες μας. Ευχαριστώ. κύριε Ανδρέασεν. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι κάπως αντίθετη σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση υποχρεώσεων και πληρωμών. Πρώτα θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιε είναι οι δυνατότητέ μα για δαπάνε και μετά να αναλαμβάνουμε τι υποχρεώσει. Θα πρέπει να ξεκινούμε ανάποδα δηλαδή. Πέρυσι το Συμβούλιο επέβαλε αυτή τη διαδικασία. Και εμεί δεν καταλάβαμε ότι αυτό θα γίνεται όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα όταν έχουμε μια κρίση. Και δεν νομίζω ότι είναι έξυπνο να μιλούμε πρώτα για υποχρεώσει. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι ότι έχουν στι τσέπε του και ποιε είναι οι υποχρεώσει πληρωμών τους. Και έτσι έρχομαι σε κάτι άλλο που ακούσαμε πολλαπλά επανειλημμένα στην Επιτροπή μας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινοτικό έλλειμμα, δεν έχει δημοσιονομικό έλλειμμα. Φυσικά δεν έχει δημοσιονομικό έλλειμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρώτα αποφασίζει τι θέλει να πληρώσει και μετά ζητά τα χρήματα από τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν ισχύει στις εθνικούς προϋπολογισμούς. Εκεί οι κυβερνήσεις πρέπει να αποφασίσουν πού θα αφιερώσουν τα κονδύλια τους και μετά προσπαθούν να βρουν ε, κονδύλια για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Δεν ζητούν απλώς να τους χρηματοδοτήσει κάποιο. Αυτοί πηγαίνουν και βρίσκουν με τα έσοδα τα φορολογικά ένα πληρώσουν τις δαπάνες που έχουν ε, αναλάβει την υποχρέωση να εκτελέσουν. πέρσι οι μικρές ομάδες δεν συμμετείχαν σε πολλές ε, διαπραγματεύσεις των προϋπολογισμών. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι αντιδημοκρατικό. Λυπάμαι κυρία Αντρέασεν, ήταν πολύ δημοκρατική η διαδικασία. Γιατί η δημοκρατία δεν σημαίνει ότι θα αποφασίζουμε με ομοφωνία αλλά ότι αποφασίσουμε με πλειοψηφία. Αυτό είναι δημοκρατία. Και όλες μας οι απόψεις ελήφθησαν με διαφανή και δημοκρατικό τρόπο. Για το σημείο αυτό, κύριε Φέρν, δύο σχόλια θα ήθελα να απευθύνω προς την κυρία Αντρέασεν. Καταρχήν, πώς διοργανώνονται οι τριμερείς διάλογοι. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα κοινοβούλια, σε όλους τους νομοθετικούς ε, τριμερείς διαλόγους μας εκπροσωπούν ο εισηγητής και ο πρόεδρος, κανείς άλλος. Και αυτό γίνεται για πρακτικούς λόγους. Δεν γίνεται ψηφοφορία, αλλά διαπραγμάτευση στον τριμερή διάλογο. Μία διαπραγμάτευση που για πρακτικούς λόγους χρειάζεται λίγους συνομιλητές. Και είναι λογικό αυτό. Είχαμε πρόβλημα πέρυσι, γιατί τότε όλοι όσοι εκπροσωπούσαν το κοινοβούλιο ήταν από την ίδια πολιτική ομάδα. Αυτό ήταν πρόβλημα, ότι όλοι προερχόνταν από μία και μόνο πολιτική ομάδα. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη αντιπροσωπευτικότητα σε ένα τριμερή διάλογο, γιατί έτσι θα μετατρέψουμε το τριμερή διάλογο σε κάτι τελείως διαφορετικό από ότι αυτό που έχει αρχικά, για το οποίο έχει αρχικά σχεδιαστεί. Η κυρία Ανδρέασεν είπε ότι πρώτα αποφασίζει για τις υποχρεώσεις και μετά ζητά κονδύλια. Λάθος. Κοιτάξτε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε ανώτατα όρια για κάθε χρόνο που είναι ανυπέρβλητα. Και έχουμε πολλά ανώτατα όρια και ανώφλια για τους ίδιους πόρους, για τις υποχρεώσεις. Αυτά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε από μόνοι μας. Είναι κοινή απόφαση όλων των κρατών μελών. Το σύστημα ιδίων πόρων έχει εγκριθεί από το σύνολο των χωρών μελών και όλες οι χώρες έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας. Μην μας λέτε τώρα ότι κάνει το κεφαλίο της η Ένωση, καταρτίζει τον προπολογισμό και μετά ζητά να τη χρηματοδοτήσουν. Αυτό δεν ευσταθεί. Ράιμερ και μετά ο James για το ίδιο θέμα. Πρώτα ο James και μετά ο Ράιμερ. Ως προς τη διαδικασία καταρχήν. Δίκιο έχεις, Ελέν. Γιατί εσύ έχεις ε, πιο μακροχρόνια πείρα από μεγάλη ομάδα από ότι εγώ από μικρή. Και συνήθως στον τριμερή διάλογο εκπροσωπείται η Επιτροπή από τον πρόεδρο και τον εισηγητή. Πολύ σωστά είπε ο Γκόραν ότι αν έχουμε περισσότερους εκπροσώπους θα γίνει πανδεμόνο στον τριμερή διάλογο. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Τώρα, υπήρξε κάποια, κάποιο πρόβλημα πέρυσι στη συνδιαλέγη για το ποιος νομιμοποιούνταν να πάει στη συνδιαλέγη. Και δεν ήταν σίγουρο ποιο μέχρι το τέλο μπορούσε να συμμετέχει. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε πού μπορούν να πάνε οι βουλευτέ και πού όχι, ώστε στο τέλος να ενημερώνεται η Επιτροπή Προπολογισμών και να λαμβάνουμε τελική απόφαση τεκμηριωμένα. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Σε ό,τι αφορά ε, το θέμα των υποχρεώσεων και των πληρωμών. Έχουμε στην αρχή υποχρεώσεις, μετά πληρωμές, αναλαμβάνουμε υπέρογγες υποχρεώσεις, δεν μπορούμε να τις χρηματοδοτήσουμε, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Και πάντα στο τέλος των δημοσιονομικών προοπτικών ε, μας λείπουν κονδύλια συνήθως συμβαίνει, αλλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, λόγω της έλλειψης χρημάτων και ρευστών που υπάρχουν στις χώρες, δεν μπορούμε να τις υποχρεώσουμε να συμβάλλουν περάνω των δυνατοτήτων τους. κύριος Μπέγκε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι για αυτές τις λήψεις αποφάσεων για θέματα υποχρώσεων και πληρωμών όπως είπαν και οι δύο προηγούμενοι, πρέπει να το συζητήσουμε κάποια στιγμή διεξοδικά για να δούμε προς τα που θα κινηθούμε, διότι έχουμε μια εξέλιξη αυτής της ε, απόκλησης που είναι όλο και μεγαλύτερη και που εν τέλει στερεί και αξιοπιστία το, τον ευρωπαϊκό ε, προϋπολογισμό. αυτά δεν είναι πολύ σοβαρά. Δεύτερο, για την διαδικασία. Υπενθυμίζω ότι Προ πολλών ετών είχαμε αντιμετωπίσει μια κατάσταση όπου και οι διαπραγματεύσει ακόμη για πολυετή ε, δημοσιονομική προοπτική Ατζέντα 2000 είχαν γίνει μοναχά από τον πρόεδρο και τον εισηγητή και μάλιστα αυτή ήταν και από την ίδια πολιτική ομάδα. Όσα ανταπάντηση μετά σε αυτό είχαμε ένα πληθωρισμό ε, ε, εκπροσώπησης στον τριμερή διάλογο. Όχι μόνο με συντονιστές αλλά και εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές και όχι μόνο ένα συνεργάτη πολιτικής ομάδας αλλά ίσως και δύο και τρεις. Ώστε να είναι τόσο πλήρης η αίθουσα από την πλευρά του Κοινοβουλίου όσο σε μια απλή διαβούλευση και αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Υπενθυμίζω και τα σχετικά με την ενημέρωση πριν από την υπόθεση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσεως που είχαμε προβλέψει ειδικά φόρμα για την εκπροσώπηση. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ώστε όλες οι πολιτικές ομάδες να διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες άλλωστε και να παρακολουθούν κιόλα ότι οι εκπρόσωποι τους πράττουν ακριβώς αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί αλλά να υπάρχει και επαρκής εμπιστοσύνη. Άρα σε ένα τριμερή διάλογο είναι καθήκον του Προέδρου της Επιτροπής ενδεχομένως και του εισηγητού να εξηγήσουν τις θέσεις τις οποίες έχουμε καταλήξει εδώ μετά από δύσκολες και κοπιαστικές συζητήσεις. Ε, κάτι το οποίο δεν γινόταν προ 10 ή 15 ετών. Υπάρχει λοιπόν η προπαρασκευή, υπάρχει και η δυνατότητα επανόδου δηλαδή να ξαναέρθουν και να εξηγήσουν τι συνέβη. Άρα με αυτόν τον τρόπο πρέπει να συνεχίσουμε χωρίς να περιοριστούν οι δυνατότητες συμμετοχής των πολιτικών ομάδων στην διαδικασία της προπαρασκευής και γνωρίζουμε ούτως ή άλλως με ποια διαδικασία ε, κατανέμονται οι εκθέσεις αλλά στον τριμερή διάλογο δεν ομιλούν εκ μέρους των ομάδων τους και παρόλο που το θέμα μου το Ταμείο Λεγγύης ξαναμπαίνει στην ημερησία διάταξη. Εγώ παρετήθηκα από το να είμαι παρόν για να μην δυσχερανθεί η εκπροσώπηση, γιατί θεωρώ ότι πρόεδρος και εισηγητής επαρκούν για να μεταφέρουν τις απόψεις μας. Ευχαριστώ αγαπητέ Ράιμερ. Συνειδητοποιώ ότι η γενεδορία του σημερινού εντό εισαγωγικών ε, του σημερινού Προέδρου είναι, δημιουργεί ε, σύγχυση. Θα προσπαθήσουμε αυτό να το χειριστούμε. Τελευταία παρατήρηση όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών και υποχρεώσεων, για να δω συνέχεια στα όσα είπε η κυρία Αντρέσεν. Προφανώ προφανώς αυτό που είναι πιο σημαντικό στο τέλος είναι τα χρήματα που θα δαπανηθούν πραγματικά. Όμω, από τη στιγμή. Με συγχωρείτε. Ε, το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε αποφασίσει να δαπανίσουμε, που έχουμε υπογράψει μια σύμβαση έργου και έχουμε προσλάβει κάποιον, έχουν γίνει τα έργα, πρέπει να τα πληρώσουμε. Και είμαστε τώρα σε μια κατάσταση που έχουμε αποφασίσει να δαπανίσουμε, η δουλειά έχει γίνει, οι υπάλληλοι έχουν προσληφθεί και τώρα λέει το Συμβούλιο, τώρα δεν έχω άλλα χρήματα. Μα αυτό είναι τρελό. Πρέπει φυσικά να διαπραγματευτούμε το επίπεδο των πιστώσεων ε, υποχρεώσεων με βάση τις δαπάνες που είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε φυσικά. Αλλά από τη στιγμή που θα έχει ληφθεί η απόφαση θα... Ε, ε, είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Και νομίζω πως πρέπει να βγούμε από αυτή την αμφισημία γιατί θα φτάσουμε σήμερα άλλη μια φορά, το επαληθεύσαμε σήμερα, θα υπάρξουν ανόητες επιπλοκές και ανεπίλητες και ερμηνεύω την σιωπή του Συμβουλίου για την παρατήρηση που έκανα ότι είμαστε στην ίδια κατάσταση όπως και τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως την πέρυσι ότι οι συνομιλητές δηλαδή που έχουμε ενώπιον μας και που λέγεται Συμβούλιο δεν είναι συνομιλητής που να έχει πολιτική εντολή για μια ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο. Στην ουσία έχουμε δηλαδή ένα συνομολητή που είναι χειροπόδαρα δεμένος από τους υπαλλήλους. Και η πολιτική που είμαστε εμείς διαπραγματευόμαστε με υπαλλήλου. Και δεν επικρίνω τους ε, υπαλλήλου. Και εγώ ήμουν υπάλληλο ε, στο Υπουργείο ε, Προϋπολογισμού. Αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει τους υπαλλήλου είναι οι πληρωμές. Είναι μια λογική λογιστική. Εμείς είμαστε όμως πολιτικοί και δυστυχώς στη διαδικασία μας δεν καταφέρνουμε να έχουμε μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων και πολιτικής φύσης διαπραγμάτευση παρά στο τέλος της διαδικασίας μετά από την ψήφο του Συμβουλίου. Και στο πρώτο εξάμεινο του έτους δεν έχουμε πραγματική ανταλλαγή απόψεων πολιτικού επίπεδου παρά τις προσπάθειές μας. Απτά, αγαπητοί συνάδελφοι, να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, αυτή την ανταλλαγή πολιτικών απόψεων που εμείς τουλάχιστον έχουμε εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμού. Και ακούσατε και την έκκληση της εισηγήτριας Φραντσέσκα Μπαλτσάνη όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις για τις οποίες θέλει να έχει τις προτάσεις όσο γίνεται πιο σύντομα ώστε να πετύχει το χρονοδιάγραμμα που μας θύμισε. Μπορούμε έτσι να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι το 6 και το 5 τα έχουμε αναβάλει. Ε, το σημείο το διορθωτικό για το 2011 Τώρα, συγκεκριμένο παράδειγμα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε δεδομένες της κατάστασης των πιστώσεων πληρωμών. Η συγγήτρια δεν μπορεί να είναι εδώ δυστυχώς. Η Σιδόνια Τζεγεύσκα γιατί αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα και ελπίζω ε, σύντομα να γίνει καλά το παιδάκι της που βρίσκεται στο νοσοκομείο και ευχόμαστε περαστικά όλοι σύσσωμοι και ότι η απουσία της ο Σαλβατόρ Γαρίγκα θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου και θα μας κάνει και μια συγκεκριμένη πρόταση. Σαλβατόρ. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο να αναπληρώσω εδώ την εισηγήτριά μας για το θέμα αυτό. Γιατί είναι ένα περίπλοκο θέμα, επίμαχο και συγκρούνται δύο διαφορετικά συμφέροντα στο θέμα αυτό. Καταρχήν το δημοσιονομικό συμφέρον που αντιστοιχεί στην Επιτροπή μας και αφετέρου το πολιτικό συμφέρον αν ικανοποιήσουμε το δημοσιονομικό συμφέρον, είπαμε συντονιστές και εξηγήσαμε σε προηγούμενες συνεδριάσεις ότι το αρνητικό αποθεματικό δεν ε, είναι αποδεκτική, εναλλακτική λύση. Και εδώ και χρόνια καταψηφίσαμε το αρνητικό αποθεματικό για τους ίδιους λόγους που το αποκηρύσουμε και σήμερα. Και δεν ήταν συνεπές να εφαρμόσουμε στην αρχή του χρόνου αρνητικό αποθεματικό ή να ζητήσουμε ένα διάταξη δαπανών στην αρχή του χρόνου προκειμένου να υλοποιήσουμε ένα στόχο που έχει δύο θεμελιώδη χαρακτηριστικά, το κατεπήγοντα χαρακτήρα και την αλληλεγγύη. Αυτά τα χαρακτηριστικά έχει το Ταμείο Αλληλεγγύης. Κατά τη γνώμη μας ήταν ε, η χαρακτηριστική περίπτωση η ιδεώδης ευκαιρία για το Συμβούλιο να τηρήσει την ε, διοργανική συμφωνία για, την, ε, για τις επαρκείς δαπάνες όταν το απαιτούσαν οι συνθήκες και ιδιαίτερα ότι υπάρχει ένας απροσδόκητος στόχος. Τι πιο απροσδόκητο από, από πιο απρόσμενο από μια θεομηνία. Ας μας εξηγήσει το Συμβούλιο. Υπάρχει κάτι πιο απρόβλεπτο από μια θεομηνία. Ας μας το εξηγήσει, επαναλαμβάνω. Υπάρχει λοιπόν ο κατεπήγον χαρακτήρας, ε, ο απρόβλεπτος χαρακτήρας και παρόλα αυτά, παρά την ανάγκη που υπάρχει και το Συμβούλιο μας εξήγησε ότι για τα 184 εκατομμύρια ευρώ χρειαζόταν νέα χρήματα. Το Συμβούλιο δεν συγκέντρωσε πλειοψηφία Οπότε προσέφυγε στο αρνητικό αποθεματικό. Από δημοσιονομική άποψη ήδη απορρίψαμε αυτή την πρόταση. Χθε όμω τον τριμερή διάλογο και παρόλο που ο Επίτροπο μα ξανά εξήγησε τι γίνεται σε τέτοιε περιπτώσει, εφαρμόζουμε δηλαδή τη θεωρία του νέου χρήματο για να ανταπεξέλθουμε στις νέε υποχρεώσει. το Συμβούλιο, η Προεδρία μα είπε ότι είναι αδύνατο να τροποποιηθεί η ή να μεταπιστούν οι ε, αντιπροσωπείς του Συμβουλίου που είναι κατά του αιτήματο αυτού που είναι κοινό και της Επιτροπής. Και μας εξήγησαν ότι στο Συμβούλιο αυτό που διακυβεύεται είναι το συμφέρον, η ευημερία και το οικονομικό μέλλον των πολιτών της ευρωπαϊκή Ένωσης που έχουν θυγεί και πληγεί σοβαρότατα από τις πλημμύρες αυτές. Και μια και χώρες αυτές που είναι η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Κροατία και η Ρουμανία αντιμετωπίζουν πολύ περίπλοκες δημοσιονομικές καταστάσεις και δυσχέρειες, χρειαζόμαστε το συντομότερο δυνατό μια κοινοτική ευρωπαϊκή λύση. Αν εφαρμόσουμε την δημοσιονομική πειθαρχία και λιτότητα και πούμε ότι απορρίπτουμε συλλήβδη την πρόταση για το αρνητικό αποθεματικό, ίσως επιτείνουμε αυτή την καθυστέρηση. Ήδη είμαστε σε δωδεκάμινη καθυστέρηση, γιατί έγιναν πέρυσι τον Απρίλιο αυτές οι πλημμύρες. Μία τέτοια λοιπόν απόρριψη θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία και οι χώρες θα καθυστερήσουν στη λήψη της κοινοτικής αντιστάθμισης και οι πλημμυροπαθείς στη λήψη της ενίσχυσης. Ο δεύτερος διορθωτικός προϋπολογισμός και πάλι μιλά για πλημμύρες και προβλέπει ένα επιπλέον κονδύλιο που αν προσθεθεί στο κονδύλιο του πρώτου διορθωτικού προϋπολογισμού μας κάνει να υπερβούμε τα 200 εκατομμύρια που είναι αυτό που προβλέπει το άρθρο 4 του Δημοσιονομικού Κανονισμού ως ανώτατο κονδύλιο για το λεγόμενο αρνητικό αποθεματικό. Οπότε η λύση που θα επιλέξουμε σήμερα θα είναι ούτως ή άλλως αποσπασματική και μερική, γιατί για το δεύτερο διορθωτικό προϋπολογισμό θα πρέπει να προστρέξουμε σε άλλη λύση, ίσως το νέο χρήμα. Αυτό είναι και το πιο λογικό δεδομένη της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά, ως εκπρόσωπος, η ε, αντικαταστάτης μάλλον της συγκίτριας ε, Συντόνιας Γέντζο εγώ θα πρέπει να λάβω υπόψη όχι μόνο την ανάγκη τη δημοσιονομική πειθαρχία και λιτότητα, αλλά λάβω υπόψη και τι πολιτικές ανάγκε. Οπότε, μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων, πιστεύω ότι θα πρέπει στην Επιτροπή μας να ψηφίσουμε υπέρ του αρνητικού αποθεματικού κατεξαίρεση. όχι όμως ανεφόρων. Δεν ξέρω αν έχετε λάβει όλοι τους όρους που προτείνουμε. Ο πιο σημαντικός όρος είναι το σημείο 2. Πέραν των στοιχείων της αιτιολογικής σκέψης, το σημείο 2 ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την επιφύλαξη του δικαιώματος πρωτοβουλίας της φυσικά, να τροποποιήσει το διορθωτικό προϋπολογισμό ε, για τα πλονάσματα για το 2010, όπως προβλέπει το άρθρο 15 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, προκειμένου να τηρηθεί αυτό το αρνητικό αποθεματικό. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να υποβάλει μία πρόταση ύψους 200 εκατομμύρων ευρώ που θα αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό των υπολείπων ε, που επιστρέφονται στα κράτη-μέλη. Έτσι, ανταποκρινόμαστε στην κατεπίγουσα κατάσταση αυτή που μας υποχρεώνει να καταβάλουμε τα 184 εκατομμύρια του Ταμείου Αλληλεγγύη συν τα 19 εκατομμύρια από το δεύτερο διορθωτικό προπολογισμό και ταυτόχρονα θα θέσουμε το Συμβούλιο ενώπιον των ευθυνών του γιατί τόσο πρόωρα προ... έβαλε το 2,9% για τους πληρωμές του 2011, κάτι που στερεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το περιθώριο λιγμών της για να τηρήσει την ανάληψη υποχρεώσεων. Όχι τις απρόβλεπτες υποχρεώσεις, αλλά ακόμη και για τις κανονικές πληρωμές των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτή είναι η πρόταση που είναι περισσότερο πολιτικής υφής παρά δημοσιονομικής, αλλά εκ μέρους της συζήτησης θα ήθελα να σας ζητήσω να υποστηρίξετε αυτή την πρόταση. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Η παρουσίαση του Σαλβάντορ ήταν πολύ ξεκάθαρη. Να προσθέσω δύο-τρεις παρατηρήσεις. Φυσικά και εκμεταλλευτήκαμε αυτή την ευκαιρία να εκφράσουμε, και το έκανα και εγώ ίδιο, να εκφράσουμε απέναντι στο Συμβούλιο την λύπη μας και την οργή μας θα έλεγα, μέχρι και την οργή μας για τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο δεν τήρησε τη δέσμευση που είχε αναλάβει το ίδιο με δική του πρωτοβουλία και που είναι τμήμα του προϋπολογισμού 2011, σύμφωνα με την οποία αν έλειπαν πιστώσεις πληρωμών και αν ήταν επίγουσα κατάσταση, θα μπορούσαν να αυξηθούν αυτές οι πιστώσεις. Αυτή είναι μια δήλωση που αρχικά ήταν μια μονομερή δήλωση του Συμβουλίου, στην οποία έπειτα συμφώνησαν και η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο και συνδεόταν με το γεγονός ότι οι πιστώσεις πληρωμών την αρχική τους ε, αύξηση την περιορίσαμε στο 2,91% και είχαμε πει ότι αν προκύψει το 2011 πρόβλημα πιστώσεων πληρωμών, το Συμβούλιο είχε αναλάβει αυτή την επίσημη δέσμευση και έθεσα την ερώτημα στο Συμβουλίο. Αν είναι αυτές οι δεσμεύσεις ε, του Συμβουλίου, θα το λάβουμε υπόψη. Θα θεωρήσουμε δηλαδή για τις μετλωτικέ διαπραγματεύσει, είτε είναι για τον ετήσιο προπολογισμό, είτε είναι για τις μασονομικές προοπτικές, ότι οι δεσμεύσεις του Συμβουλίου δεν ισχύουν, δεν αξίζουν τίποτα. Και μάλιστα ρώτησα, από τη στιγμή που, όπως εξήγησε ο Σαλβατόρ Γκαρίγκα, αυτή η ευκολία για αρνητικό απόθεμα εξαντληθεί με μια 200 εκατομμύρια ευρώ με μια. Τι θα κάνετε αν σε λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες βρεθείτε ενώπιον απρόσμενων δαπανών που όμως κριθούν απαραίτητες. Ποια θα είναι η θέση του Συμβουλίου και εκεί. Δεν λάβαμε απάντηση από πλευρά του Συμβουλίου. Τώρα, έχουμε Ενώπιον αυτού του προβλήματος για το οποίο ήδη έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες συνεδριάσεις, επί χάρτου υπάρχουν τρεις διαφορετικές επιλογές. την απορρίπτουμε, πράγμα το οποίο άμεσα θα οδηγούσε σε συνδιαλλαγή. Υπάρχει η δυνατότητα της μη αντίδρασης και εκεί μέσα σε μια χρονική περίοδο έξι εβδομάδων αν δεν απαντήσει το κοινοβούλιο η στάση του Συμβουλίου είναι, εγκρίνεται αυτόματα και έπειτα υπάρχει και αυτό που προτείνει ο εισηγητής που λέει δεδομένες της φύσης του προβλήματος Δηλαδή θέλουμε να βοηθήσουμε πληθασμούς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και που περιμένουν ήδη εδώ και πολλούς μήνες. Είναι δύσκολο να μην δοθεί συμφωνή γνώμη και μάλιστα γρήγορα. Αν επιλέγαμε να μην ψηφίσουμε, θα καθυστερούσαμε ακόμα για έξι εβδομάδες την εφαρμογή, την απελευθέρωση των ε, πιστώσεων, για για, για τις οποίες υπάρχει μάλλον μεγάλη συνένεση μέσα στο Κοινοβούλιο και, και στο Συμβούλιο για να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο Σταθεροποίησης για τα ποσά αυτά και για με τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά για να υπογραμμίσουμε τη διαφωνία μας με τη θέση του Συμβουλίου προτείνεται σε αυτή την προφορική τροπολογία που παρουσίασε ο Σαλβαντόρ να, να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ο σεβασμό στην ε, ε, δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλία, τα χρήματα στο τέλος του έτους να αντιστοιχούν σε ένα αντίστοιχο πλεόνασμα εκτέλεσης. Γιατί το αρνητικό απόθεμα σημαίνει να στείλουμε στο τέλος της χρονιάς την επιλογή χρηματοδότησης που δεν έχουμε το θάρρος να κάνουμε τώρα. Αυτό γίνεται στην ουσία. Αυτή η δυνατότητα, αυτό το τρίκ, αυτή η τεχνική να το αναβάλουμε για αργότερα περιορίζεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Σε ένα μόνο θέμα, σε ένα μόνο φάκελο εξαντλείται αυτό το απόθεμα. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν με τον εισηγητή είναι να ανακοινώσουμε εκ των προτέρων ότι η θέση μας για το τέλος του χρόνου είναι ότι πρέπει αυτό να χρηματοδοτηθεί όχι με αναδίπλωση αλλά με τη χρήση των των εκτέλεσης. Με όλο το σεβασμό στους όρους της Κομισιόν τι σημαίνει ότι προτείνουμε μια συγκεκριμένη διατύπωση αλλά φυσικά αν η Κομισιόν δεχτεί την αρχή αλλά έχει μια κάποια διαφορετική διατύπωση, αυτό είναι τα δική της ευθύνη. Λοιπόν, ο Γκέραντα Φέρμα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο γιατί συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο ομιλητή για το πώς πρέπει να το χειριστούμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φανεί ενωμένο και παρά Παρ' όλα αυτά θέλω να κάνω κάποια σχόλια. Δεν είναι καλή λύση. Δεν είναι διαφανής, απλώς αναβάλει το πρόβλημα. Είναι καλό λοιπόν τώρα να κάνουμε κάποιες τροπολογίες ε, όπου να επικρίνουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είμαι πολύ απογοητευμένος για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το Συμβούλιο αυτό το θέμα. Με τελείω αντιφατικό πνεύμα σε σχέση με την κοινή δήλωση που κάναμε πέρυσι. Είναι τελείω αντίθετο. Και θα είναι πρόκληση για τις σχέσεις μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων όπως είπατε, είναι απλώς μια καθυστέρηση. Είναι ένα πολύ ορατό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πληρώνει για τις καταστροφές μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης. Αφορά την ίδια την ιστεροφημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε όμως ωστόσο επιλογή από το να ακολουθήσουμε την σύσταση του εισηγητή. Έχω μια ερώτηση στο Ράιμερ Μπέγκε για το δικό του κομμάτι αυτής της πρότασης, τροπολογίες 2, 3 και 4, τις οποίες κατέθεσε πριν να, να τεθεί επιτάπητος αυτή η λύση, τις χρειαζόμαστε ακόμα, γιατί εγώ θεωρούσα πως ε, σχετίζονταν περισσότερο με την προηγούμενη κατάσταση του αρνητικού, δηλαδή αποθεματικού. Αλλά δεν ξέρω. Ίσως να ισχύουν ακόμα. Απλώς μια ερώτηση κάνω. Μάλιστα, θα μας απαντήσει ο Ράιμερ. Και όσο το σκέφτεται, να δώσω το λόγο στον Λάζλο Σούριαν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εσείς μας παρουσιάσετε τρεις εναλλακτικέ λύσεις και μία από αυτές είναι να απορρίψουμε αυτή την κακή λύση, γιατί από δημοσιονομική άποψη είναι κακή αυτή η λύση. Γιατί από πολιτική άποψη μπορεί να είναι εφικτή, αλλά είναι απαράδεκτο για την εικόνα, για την έγκλη και το κύριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κυλιδώνει την ίδια την υπόλοιψή μας. Μία άλλη πιθανή λύση είναι να απόσχουμε, ώστε με την σιωπηρή μας συνένεση να αφήσουμε να τεθεί σε ισχύ η πρόταση του Συμβουλίου. Αλλά και αυτό θα δώσει μια κακή εντύπωση για μας, γιατί δίνει την εντύπωση ότι συμφωνούμε για κάτι με το οποίο στην ουσία διαφωνούμε. Οπότε η μόνη λύση που μας απομένει και είναι το μη χείρον, είναι να δεχτούμε την πρώτη τροπολογία και το Κοινοβούλιο να το δεχτεί. Έτσι εκφράζουμε και τη γνώμη μας στο κείμενο. Αλλά έχω και μια γενικότερη παρατήρηση. Νομίζω ότι καλό είναι να έχουμε μια καλύτερη εικόνα εκ των προτέρων, γιατί πολλές πληρωμές εξαρτώνται από τις τιμές της αγοράς. Αλλά το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης και το Ταμείο Ελληνικής δεν μπορούμε να τα προσδιορίζουμε εκ των προτέρων πόσα κονδύλια θα χρειαστούν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εκ των προτέρων πόσες πυρκαγιές θα λάβουν χώρα ή πόσες ε, ε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή θεομηνίες ή πλημμύρες, ούτε πόσοι θα είναι οι πληγέντες, ούτε πόσες χώρες θα πληγούν. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό εκ των προτέρων για το Ταμείο Αλληλεγγύη. Γι' αυτό και στο Ταμείο Αλληλεγγύη ισχύουν διαφορετικοί κανόνε. Στη Γεωργία, στο Γεωργικό Ταμείο, προβλέπουμε πολύ ψηλότερα κονδύλια από τα αρχικά, ώστε να υπάρχει ένα περιθώριο λιγμό και μετά τα υπόλοιπα τα επιστρέφουμε στα κράτη-μέλη. Αλλά για τι περιπτώσει αυτέ όταν δημιουργήθηκαν αυτά τα ταμεία, δεν προβλέφθηκε αυτή η δυνατότητα για το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση και αλληλεγγύη και δημιουργούνται πολύ τεταμένες συζητήσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Οπότε όταν ε, μιλούμε για τα θέματα αυτά θα πρέπει προηγουμένως να δούμε πώς ε, υπολογίζουμε τις πιστώσεις πληρωμών και να κάνουμε και μια γενική συζήτηση για τα δύο ταμεία. Γιατί δεν έχουμε αρχικά πιστώσεις πληρωμών ενός εκατομμυρίου στις αρχές του έτους, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι δαπάνες ε, και να κάνουμε μια αναδιάταξη προς το τέλος του έτους. Έχουμε μικρές ε, ποσότητες από την αρχή, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο και αυτό δημιουργεί πολύ αρνητική εντύπωση για μας στους Ευρωπαίους πολίτες. Η ε, κυρία Ανδρέασεν, ευχαριστώ. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί θα πρέπει σώνει και καλά να λάβουμε την απόφαση σήμερα. Ούτως ή άλλως οι πλημμύρες έγιναν πριν από ένα χρόνο. Γιατί δεν περιμένουμε ε, και τον δεύτερο διορθωτικό προϋπολογισμό και μετά, ανάλογα με το τι θα αποφασίσουμε και για το δεύτερο διορθωτικό προϋπολογισμό, να επανέλθουμε και σε αυτό το θέμα. Είναι θέμα λίγων εβδομάδων ούτως ή άλλως. Και θα αποφύγουμε και τη χρήση του αρνητικού αποθεματικού που από άποψη είναι πραγματικά κάτι τελείως παράλογο και παράδοξο. Ευχαριστώ. Καλά, καλώς το θέτετε. Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα και το συζητήσαμε και την περασμένη φορά. Αλλά έχουμε τέτοια καθυστέρηση που όντω θα μπορούσαμε να περιμένουμε ακόμη λίγε εβδομάδε. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε καθυστερήσει υπερβολικά, γιατί η αρχική καθυστέρηση οφειλόταν ίσω στι διοικητικέ αδυναμίες των ε, ενδιαφερόμενων χωρών. Μετά καθυστέρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθυστέρησε και το Συμβούλιο και ήρθαμε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Γιατί αν τώρα πούμε όχι και καθυστερήσουμε ακόμα περισσότερο, θα φανούμε εμεί ω ε, οι κακοί μαθητέ, το Κοινοβούλιο δηλαδή, ενώ εμεί προσπαθήσαμε από την αρχή να είμαστε άψογοι και υποδειγματικοί. Όπω είπε η συγγήτρια, θέλουμε να αποζημιώσουμε ουσιαστικά κάποιες τοπικές αρχές, ε, ε, εθνικές διοικήσεις ή ιδιώτες ή κάποιες επιχειρήσεις που αποζημίωσαν ε, ή μάλλον που διόρθωσαν τις ζημίες που ενέσκεψαν εξαιτίας των θεμηνιών. Ουσιαστικά με την πρόταση αυτή βοηθούμε τους εθνικούς ή τοπικούς προϋπολογισμούς των χωρών που βοηθούμε. Αυτό το στόχο έχει και το Ταμείο της Ελληνικής η ενίσχυση του Ταμείου Ελληνικής ουσιαστικά εξυπηρετεί τη δημόσια διοίκηση σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Η κυρία Βέρτμαν ζήτησε το λόγο. Κόσλικ. Και μετά θα δώσω το λόγο στο Ράιμερ για να απαντήσει την ερώτηση που το έκανε ο Γκέραν Φέρ. Η κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν σας κατάλαβα καλά, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πληγέντες. Το θέμα είναι με τι κονδύλια, από πού θα προέρθουν αυτά τα κονδύλια, από ποιο σημείο του κοινοτικού προπολογισμού. και έχω και κάποιες αντιρρήσεις. Φυσικά έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες, απέναντι στους συμπολίτε μας. Και θα πρέπει να δράσουμε αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας. Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως θα πρέπει να αποφασίσουμε από κοινού από πού θα προέλθουν αυτά τα κονδύλια. Έχω και μία παρατήρηση ως προς την τροπολογία 1. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή. Εντάξει, προσοχή, έκκληση. Αλλά θα ήθελα να είμαστε πιο κατηγορηματικοί, δεν ξέρω αν, είναι αν υπάρχει πρόβλημα με τη γερμανική μετάφραση, γιατί δεν υπάρχει κάτι υποχρεωτικό. Δεν αρκεί μια απλή έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να υποχρεούται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φτάσουν ε, τα κονδύλια αυτά στου πλημμυροπαθεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόσλικ. Ευχαριστώ. Μιλούμε για ένα μείζον πολιτικό ζήτημα εδώ. Προτείνεται μια λύση και νομίζω θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις διάφορες χώρες μεταφέρουν τις συζητήσεις που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς το συντομότερο δυνατό, μετά τις ε, καθυστερήσεις της τεράστιες που έγιναν ήδη, πώς θα φτάσουν τα χρήματα στους πληγέντες. Δεν θα πρέπει να παρατείνουμε ακόμη περισσότερο αυτή την καθυστέρηση και μάλιστα να φανούμε εμείς ως υπέτη της καθυστέρησης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί ο απλός πολίτης δεν παρακολουθεί όλη την περίπλοκη συζήτηση για τον προπολογισμό του 2012. Αυτό που βλέπει ο απλός πολίτης είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν πήραν ακόμη τα χρήματα που δικαιούνται. Όντω αυτό που είπε πριν και ο Λάζλο Σούριαν για τους Ούγγρους. Ράιμερ, θες να απαντήσει στην ερώτηση του Γκέρον. Äh, Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο Σαλβαντόρ όσον αφορά τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου και λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τα όσα μας είπε. Όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης, εγώ θα ήθελα απλώς να πω ότι το, η τροπολογία 1 ε, είναι κάτι που δεν έχει και πολύ νόημα γιατί η Κομισιόν ούτως ή άλλως έχει υποχρέωση να επαληθεύει. Ε, άρα λοιπόν η αλλω εχει την υποχρεωση κατέστη περιττή. Για τα 2, 3 και το 3 θα τα άφηνα. Ο να έχει δίκιο, αλλά για το 4 χρειάζεται μια αλλαγή περιμένοντας ε, την, απάντηση, την θέση του Συμβουλίου θα πρέπει να αφαιρεθεί εκεί που λέει Waiting ε, Council Position. Αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί, αλλά το τέλος θα πρέπει να παραμείνει γιατί έχει σχέση και με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Ώστε να καταλάβουν όλοι ποια είναι τα προβλήματα τα οποία μας απασχολούν. και για τη μελλοντική χρήση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Πρόεδρε, θα ήθελα άλλη μια φορά να πω το εξής. το Συμβούλιο χωρίς να περιμένει την έκβαση του του διαλόγου προέβησε ανακοινώσεις με παράξενο τρόπο, χωρίς να σέβεται, χωρίς να σεβαστεί τα χρονοδιαγράμματα, τα τεχνικά και γι' αυτό και βρισκόμαστε και μέσα σε μια δύσκολη θέση ε, και άρα και θα αντιδράσουμε με κάπως ασυνήθιστο τρόπο και εμείς γιατί η διαδικασία που ακολούθησε το Συμβούλιο παραβιάζει την κανονική διαδικασία. Άρα λοιπόν δεν ε, ε, ενήργησε μέσα στο ευρωπαϊκό πνεύμα συνεργασίας με τα άλλα θεσμικά όργανα το Συμβούλιο και ίσως το Συμβούλιο να μην έχει οριμάσει για να διαλλαχθεί σωστά με το Κοινοβούλιο. Έχετε δίκιο και ο Γκέραν έχει δίκιο και εγώ το είπα για να διαμαρτυρηθώ απέναντι στο Συμβούλιο ότι δεν επικράτησε η καλή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων ε, για την οποία όλοι μας έχουμε δεσμευθεί. Από τη στιγμή όπου έχουμε έναν τριμερή διάλογο όπου έχουμε γράψει το θέμα στην ημερήσια διάταξη, το μήνυμο ευγένεια ε, θα σήμαινε ότι θα περιμένουμε το τέλος αυτού του τριλόγου πριν να λάβουμε θέση. Ενώ το Συμβούλιο έλαβε θέση στις 15 Μαρτίου, δύο εβδομάδες πριν το διάλογο. Το οποίου η ημερομηνία ήταν γνωστή και το περιεχόμενο γνωστό. Εγώ διαμαρτυρήθηκα. Είναι πολύ άσχημη συμπεριφορά και ελπίζω το Συμβούλιο να το λάβει υπόψη, τη διαμαρτυρία μου. Ο Κέραν θέλει να αντιδράσει στην απάντηση του Ράιμερ. Να νομίζω πως βασικά είναι εντάξει, αλλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για την τροπολογία 2 και 3 αυτό ισχύει μόνο για τις πληρωμές και όχι για τις ε, υποχρεώσεις. Γιατί βάλαμε λοιπόν τη λέξη υποχρεώσεις στην τροπολογία 3, αφού έχει να κάνει μόνο με τις πληρωμές. Θα πρέπει να διαγραφεί η λέξη ε, υποχρεώσεις στην τροπολογία 3, αν δεν κάνω λάθος. got nothing to do with commitments. Mm-hmm. On peut se passer du mot commitments. Όντως. Μπορεί όντω να διαγραφεί η λέξη commitments. No, αν μου επιτρέπετε να πω ότι το Ταμείο Λεγγύης κινητοποιείται μόνο για ανάγκες άνω των ε, ανοφλίων για τις υποχρεώσεις. Γι' αυτό λοιπόν αυτό αναφέρεται στην ειδική δομή του Ταμείου Αλληλεγγύης. Ναι, κατάλαβα ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης λειτουργεί για υποχρεώσεις και πληρωμές ταυτόχρονα και η απόφαση του Συμβουλίου είναι να δεχτούμε τις ε, υποχρεώσεις και για τις πληρωμές να τις δεχτούμε και αυτές αλλά με την προπόθεση ότι θα χρηματοδοτηθούν από το αρνητικό αποθεματικό και άρα δεν είναι αφύσικο να αναφέρουμε υποχρεώσεις και πληρωμές στην τροπολογία μας. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Pardon. À Για πάρτε αναχείρες τον κατάλογο ψηφοφορία και καταρχήν θα ψηφίσουμε για την έκθεση της Ιδόνιας και μια σειρά τροπολογίες προφορικές που παρουσίασε ο εισηγητής και ο πρόεδρος της Επιτροπής προπολογισμών, όπως μας εξήγησε ο Σαλβαντόρ. Λοιπόν, να ψηφίσουμε ένα μπλοκ τις τροπολογίες που αφορούν τα εκτιμώντας, τα, τις τέσσερις πρώτες δηλαδή, υπέρ, κατά, δύο, αποχές, μία αποχή, μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την ε, συνδυαστική προφορική, την προφορική συνδυαστική του εισηγητή, που είναι το κείμενο με την περισσότερη ουσία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, δύο. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 1, Herzog δεν καταπίπτει, αλλά ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Οι σοσιαλιστές. Που είναι πολύ περιορισμένοι, σε ποιότητα, αλλά σε ποσότητα. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Δεν εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Και έχουμε την τροπολογία στην παραγραφό 3. Εδώ είναι μια διευκρίνηση τεχνική σχεδόν φύση. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, Αποχέ. μία, εγκρίνεται. Επίσης. Τελική ψηφοφορία γιατί είναι διορθωτικός προπολογισμό. Ποιοι είναι υπέρ του διορθωτικού προπολογισμού. Ο Λάζλο Σουριάν είναι υπέρ. Κατά. Δύο. Αποχές. Μία αποχή. Μάλιστα. Διορθωτικός προπολογισμό υπαριθμών 1 εγκρίνεται λοιπόν με... Η απόφαση εγκρίνεται και τώρα περνάμε στην έκθεση του Ράιμερ Μπέγκερ για την απόφαση κινητοποίηση για το Ταμείο. Τώρα που έχουμε τους διαθέσιμους τους πόρους μπορούμε να αποφασίσουμε και να τους χρησιμοποιήσουμε για την εφαρμογή και τη λειτουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης υπέρ των δύο εν λόγω χωρών. Τροπολογία χέρια. Ο Ρέμερ μας εξήγησε ότι ήταν κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία εποχή. Περίπτωση. Τροπολογίες 2 και 3. Unblock. Υπέρ. Κατά. Ο Γκέραν απλώς κουνάει το κεφάλι του. Αποχές. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Τροπολογία 4. Με μια προφορική τροπολογία. Εκεί δηλαδή θα καταργήσουμε το waiting house position, γιατί έχουμε τη θέση του Συμβουλίου υπέρ, κατά Ένα αποχέ, μία αποχή. Ευχαριστώ. Τελική ψηφοφορία για αυτή την απόφαση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και μία αποχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και την εισηγήτρια και τον αντικαταστάτη της. Nous revenons maintenant à notre ordre du jour et euh, au titre des donc nous Επανερχόμαστε στην ημερήσια διάταξη. Σημείο 11. Ψηφοφορίες πάλι. Έκθεση Γένσεν. Απουσιάζει η κυρία Γένσεν, αλλά την αντικαθιστά ο κύριος Χάγκλουντ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ εξ ονόματος της κυρίας Γένσεν τους συναδέλφους για τις 18 τροπολογίες που κατέθεσαν. Η κυρία Γένσεν τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι πολιτικές αυτές για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Βέβαια με το μηχανισμό αυτό τίθεται ορισμένα προβλήματα που ακόμα δεν έχουν αντιμετωπιστεί όπως θα έπρεπε. Συμφωνεί ότι χρειάζεται να ενισχυθεί ε, το κείμενο για την ε, ανάληψη ευθύνης των υπολόγων στις χώρες να περιληφθεί και το EDF στο νέο προϋπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και να σημαίνει, σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα χρήματα συνολικά για την ανάπτυξη και αυτό που θέλω να σας μεταφέρω αυτά είναι που ήθελα να σας μεταφέρω μάλλον και είμαι έτοιμος αν θέλετε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ο πρόεδρος σας ευχαριστώ, ο Γιώργος Φέρμα. Πολύ σύντομα. Οι προτάσει τη εισηγήτρια είναι καλέ. Έχουμε καταθέσει ορισμένε τροπολογίε ενισχυτικέ του κειμένου. Έχει προταθεί ψηφοφορία κατά τμήματα στην τροπολογία 2 για να διαγραφεί μια φράση στη μέση τη τροπολογίας μα. Εγώ είμαι διατεθειμένο να αποσύρω τη συγκεκριμένη αυτή φράση, ώστε να μην χρειαστεί ψηφοφορία κατά τμήματα γιατί συμφωνώ και εγώ ότι μπορεί να προκαλέσει κάποια παρανόηση η διατύπωση. Αποσύρω λοιπόν το τμήμα που επιθυμεί να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία η κυρία Γένσεν. Κατά τα άλλα θα είμαστε υπέρ. Τώρα για την τροπολογία 17. Εκεί έχω μία ερώτηση προς την εισηγήτρια. Ίσως όμως να έχει εξηγήσει τον κύριο Χάγκροντ γιατί είναι απούσα. Αντιδρά στην προκλητική διατύπωση της πρώτης φράσης που ε, λέει ότι η διεθνή κοινή γνώμη θεωρεί την Ευρώπη ακόμα έναν οικονομικό γίγαντα αλλά πολιτικό νάνο. Ε, αυτό είναι αληθές, έστω και αν φαίνεται προκλητικό. Ε, είμαστε διτεθειμένοι να αποσύρουμε και αυτό το τμήμα. Αλλά το δεύτερο τμήμα τη τροπολογία αυτή είναι σημαντικό και πρέπει να υπερψηφιστεί. Εάν αυτό διευκολύνει την εισηγήτρια να βάλει ένα συν, τότε είμαστε διατηθειμένοι να αποσύρουμε το πρώτο αυτό μέρο, έστω και αν εμένουμε στην αλήθεια τη δήλωση να μην εμφανιστούμε και αγενείς απέναντι στην κυρία Άστον, λέει ο πρόεδρος. Ε, η κυρία Χάγκλουντ. Κύριε. Κύριε Χάγκλουντ. Η πρώτη φράση αυτή θεώρησε ότι είναι κατάλληλη για τη γνωμοδότηση. Αν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ψηφοφορία κατά τμήματα ε, και μετά από την λέξη νάνος ε, να κάνουμε εκεί το χωρισμό δηλαδή και να είμαστε υπέρ του δεύτερου τμήματο. Μάλιστα, καλά. Σας ευχαριστώ. Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία λοιπόν. Τροπολογία 1. Εισηγείται αντίθετη, υπέρ. Κατά. Α, νομίζω πρέπει να γίνει καταμέτρηση. Θα πρέπει να γίνει καταμέτρηση. Έχετε τις κάρτες σας για να γίνει τότε ονομαστική ψηφοφορία. Δεν έχω την κάρτα μου του κ. Σπόρτας. Α, δεν λειτουργεί ούτως ή άλλως το μηχάνημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Α, λειτουργεί, λειτουργεί. Καλά. Ε, πάρτε τις κάρτες σας. Δύο κακοί μαθητές, Πόρτας και εγώ, δεν έχουμε τις κάρτες μας. Α, τρεις κακοί μαθητές. Ο κ. Θα προσπαθήσουμε πάντως. Αρχίζει η ψηφοφορία. Βάλτε την σωστά όμως. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Ψήφι 14 υπέρ, 11 κατά. Ο κύριος Πόρτος απέχει. Εγκρίνεται λοιπόν γιατί υπάρχουν και δύο ακόμη ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 2 εδώ δεν ζητείτε πια ψυχοβαρή τμήματα γιατί αποσύρεται το τελευταίο μέρος της φράσης. Ψήφοι υπέρ. Κατά. Τρεις κατά. Αποχές. Χωρίς αποχές. Εγκρίνεται. Η τρία του κυρίου Πόρτας. Η συγκέντρια αντίθετη. Ψήφι υπέρ του κ. Πόρτος. Κατά. Αποχές. Μια αποχή, μια αποχή. Απορρίπτεται. Τέσσερα του Ιόραν Φάρμ. Πρώτα, μια τροπολογία προφορική, εκεί που λέει in this regard, εν προκειμένου. Υποθέτω ότι όλοι είστε υπέρ. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, Βάζουμε λοιπόν την φράση αυτή εγκρίθηκε. Για το υπόλοιπο παραμένει χωρισμένη σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα εισηγείται είναι υπέρ, ψήφι υπέρ. Το πρώτο τμήμα της 4, κύριε Χάκλουντ. Είστε υπέρ, ε. Καλά, εισηγείται λοιπόν υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν το δεύτερο τμήμα, εκεί που λέει υπογραμμίζει ό,τι κλπ, εκεί εισηγείται η αντίθετη ψήφι υπέρ. Κατά η αριστερά. Οι υπόλοιποι. Μία αποχή. Απορρίπτεται λοιπόν το δεύτερο μέρος. Τροπολογία 5 της κυρίας Ανδρέασεν. Εισηγείται η αντίθετη ψήφι υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έξι Πόρτας. Η συγγήτρια είναι κατά. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ευχαριστώ. Απορρίπτεται. Έπτα του κυρίου Μπέργκε η συγκεντριά είναι αντίθετη, υπέρ. απομονωμένο σύνορα η και σήμερα. Με ωστόσο την ενθουσιώδη υποστήριξη των κυρίων Ανδρέασεν και Βέρτμαν. Κατά σχόλιο του Πρόεδρου. Ευχαριστώ. Αποχές. Παρά την ενθουσιώδη υποστήριξη ορισμένων ε, ευρωβουλευτών, Ιτήθη ωστόσο η τροπολογία του κ. Μπέογε. 8. Κοσλόφσκι. Προφορική τροπολογία του εισηγητού που προτείνει το κείμενο αυτό να προσθεθεί στην παράγραφο 4β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και ομόφωνα μάλιστα. 9. Πάλι του κ. Κοσλόφσκι. Εισηγείται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 πόρτας εισηγήτρια αντίθετη υπέρ κατά αποχές μεγάλη η πλειοψηφία των αντιθέτων ε, ε, απορρίπτεται λοιπόν της κυρίας Αντρεάσεν η 11 υπέρ βλέπω 5 κατά αποχές απορρίπτεται 12 του κ. Πόρτας υπέρ έξι κατά άνω των έξι αποχές απορρίπτεται πάλι όμως με ασυνήθιες πλειοψηφίες 13 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 14 της κυρίας Ανδρέασεν. Η συγκίτρια είναι αντίθετη υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 πόρτας. Η συγκίτρια αντίθετη υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 16 φαν υπέρ εισηγητρία ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 17 Γιώραν αν κατάλαβα αφαιρείτε τη φράση περί γίγαντος και νάνου δεν χρειάζεται άλλα ψηφοφορία κατά τμήματα αφού εξαφανίστηκαν οι γίγαντες νάνοι τα υπόλοιπα ε, βρίσκουν την ισχύτητα σύμφωνη. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκρίνεται η 17. 18. Φαρμ. Συγχαρητήρια είναι αντίθετη. Ψήφι υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Στο σύνολό της η τροποποιημένη ε, έκθεση υπέρ, κατά, τρεις κατά αποχές, χωρίς αποχές, εγκρίνεται και συγχαίρω την εισηγήτρια και τον κύριο Χάγκλουντ που την αντικατέστησε. Και τώρα έχουμε μια έκθεση του ίδιου του κύριου Χάγκλουντ για την ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου, ε, ε επανεξέταση μάλλον, του 7ου προγράμματος πλαισίου έρευνας. Ο ίδιος διευθυντής έχει κάποια παρατήρηση. Όχι, θα ευχαριστήσω μόνο τους σκιώδης ηγητές για την επικοδομητική συνεργασία και μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως στην ψηφοφορία, εάν συμφωνείτε. Καλά. Τροπολογία 1. Αυτή έχει αποσυρθεί, αν ε, τα βλέπω καλά. Δύο, Κλούτε Πόρτας, εισηγητής αντίθετο. υπέρ, η αριστερά υπέρ, με συγχωρείτε, Τέσσερι ενώρο κατά, Αποχέ. απορρίπτεται. Τρία, βον, εισηγητής υπέρ, ψηφί υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Τέσσερα του ίδιου εισηγητού του ίδιου καταθέτοντος δηλαδή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική α κεφαλαίο του εισηγητού ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 και 6 επομένως εκπίπτουν 7 κλούτε εισηγητής αντίθετος ψήφι υπέρ ψήφι αριστερά, αλλά δεν είναι πολύ άριθμη. Κατά αποχές απορρίπτεται. οκτώ του κ. Χάγκλουντ. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. εννέα βόν. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. δέκα Καρβάγιο συγκριτής υπέρ ψήφι ε, της κυρίας Καρβάλιο ναι. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 λαβία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 βον εισηγητής υπέρ ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή προφορική τροπολογία υπάρχει μόνο ένα του εισηγητού προτείνω μόνο τις λέξεις project partners αυτή, αυτή είναι το νόημα αυτό είναι το νόημα της ε, τροπολογίας υποστήριξη για να βρεθούν ε, εταίροι στην αλλαγή του έργου. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 των κ. Κρούτε και άλλων. Εδώ ο εισηγητής έχει προτείνει προφορική τροπολογία. Κ. Πόρτας. Τα προγράμματα των χωρών μελών. Μια μικρή προσθήκη δηλαδή που έχει μάλλον τεχνικό χαρακτήρα. Συμβάλλει στην κατανόηση του κειμένου. Ψηφίζουμε λοιπόν με αυτήν την ε, προφορική διευκρίνηση. Ψήφι ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 της κυρίας Καρβαγιού και του Σαλβαδόρ Γαρίγα. Συγητής υπέρ, ψήφι υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 15 των ιδίων. Εισηγητής υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 16 κλούτε. Εισηγητής υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον ο εισηγητής ήταν κατά. Απορρίπτεται λοιπόν το εδώ. Τελική ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά αποχές δύο ψήφοι μία αποχή ευχαριστώ τον εισηγητή του οποίου η έκθεση εγκρίνεται συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι καλά λοιπόν θα προχωρήσουμε τότε στην μεταφορά στις, στα εμβάσματα τη 13 λείπει η εισηγητή, ο Σαλβαδόρ είναι σε θέση να εξηγήσει τις μεταφορές. Για τις μεταφορές πιστώσεων, Σαλβαδόρ. Μήπως θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε. Ah, C'est ça. Euh, sur les virements 6 et 8 για τις μεταφορές 6 και 8 γιατί η συγγήτρια δεν θέλει να εξετάσουμε τη μεταφορά πιστώσεων 7 για τις μεταφορές 6 και 8 πρόκειται για το αποθεματικό κατεπίγουσας ενίσχυσης θέλουμε ενεργοποίηση της κατεπίγουσας ενίσχυσης γι' αυτό και απαιτούνται κάποιες μεταφορές πιστώσεων και αυτό γίνεται για την ανθρωπιστική δράση σε χώρες που επλήγησαν από θεομηνίες ή άλλες καταστροφές. Σαλβαντόρ. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τις προτινόμενες μεταφορές πιστώσεων. Η εισηγήτρια προτείνει να τις υπερψηφίσουμε. Ωραία. Θα βοηθήσουμε ουσιαστικά τα θύματα του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη και την ακτή του του. Ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ. Je vous remercie. Contre. Κατά. Αποχές. Ωραία, εγκρίνονται οι δύο μεταφορές πιστώσεων. Ευχαριστούμε, Σερβαντόρ. il ne nous reste plus μας έμεινα τώρα το σημείο 8 καταρχήν, αλλά απουσιάζει ο κύριος Κάλφη. Οι σοσιαλιστές απουσιάζουν γενικώ, οπότε δύσκολα θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων. Ερήμην του εισηγητού. Έχετε λάβει το σχέδιο έκθεσης. Γνωμοδότηση μάλλον. Αν έχετε σχόλια προς τον εισηγητή, μπορείτε να το τα μεταβιβάσετε ίσως και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το σημείο 15 έχει αναβληθεί της κυρίας Μόνικα Ολμάιερ. Οπότε εξαντλήσαμε την ημερήσια μας διάταξη. Άρα να σας κοινοποιήσω την ε, ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης που θα είναι 13 και 14 Απριλίου. Είναι πολύ σημαντική η συνεδρίαση της 13ης Απριλίου γιατί θα συναντηθούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια με θέμα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το συντονισμό κοινοτικού προϋπολογισμού με τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ να μείνουν στην αίθουσα οι συντονιστές γιατί μας απέμεινε λίγος χρόνος οπότε ας αξιοποιήσουμε και τη διερμηνία. Και ευχαριστώ και τους διερμηνείς που θα παραμείνουν στη συνεδρίαση. Λύεται η τακτική συνεδρίαση τη Επιτροπή.